Buenas tardes. Buenas tardes a todos y si les parece vamos a comenzar. Καλό σας απόγευμα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση σας παρακαλώ αν συμφωνείτε. Vamos a comenzar. Να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας. Καταρχήν, έχουμε την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Γνωρίζετε ότι εφόσον το ζήτησαν ορισμένοι βουλευτές, θα τροποποιήσουμε την ημερησία διάταξη. Θα έχουμε μια μικρή αλλαγή. Το σημείο 5 του κυρίου Ρωμέβα σε σχέση με το σχέδιο ανασύστασης του αριθρού τόνου θα το δούμε την Τετάρτη ως σημείο παριθμό 18. Συμφωνεί. Αυτή είναι η μόνη πραγματική τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης και επίσης ε, να σας πω ότι έχουμε και web streaming αυτής της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατηρήση για την ημερησία διάταξη, να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Λοιπόν, εγκρίνουμε και τα πρακτικά τη συνεδρίαση 24η ω 26η Ιανουαρίου ω ε, ήθιστε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνονται. Σημείο 3, ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν ε, έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα να σα αναφέρω και να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, την κοινή ελευτική πολιτική σε σχέση με το βασικό κανονισμό. Έχουμε υλοποιήσει διαδοχικές συνεδριάσεις για το θέμα αυτό και σήμερα τι θα κάνουμε. Θα ακούσουμε την εισηγήτρια η οποία θα παρουσιάσει τα εγγραφά εργασίας χωρίς χρονοτριβή λοιπόν. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρόντουστ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε για το βασικό κανονισμό με έγγραφο εργασίας. Βέβαια, είναι ατυχής η συγκυρία γιατί λείπουν πολλοί συνάδελφοι. Ελπίζω να έρθουν αργότερα κάποιοι ακόμη. Τους προηγούμενους μήνες μιλήσαμε εντατικά για διάφορες πτυχές της κοινή αλληλευτικής πολιτικής Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε γενικότερα το θέμα της μεταρρύθμισης και να συνδυάσουμε τα επιμέρους θέματα και άξονες μεταξύ τους. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους για την καλή σας συνεργασία. Τονίζω ότι το έγγραφο εργασίας μου αποτελεί βάση για συζήτηση και ρητά λέω εδώ ότι περιμένω με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας και θέλω να συμπεριλάβω όσο γίνεται περισσότερες παρατηρήσεις σας. Επειδή είναι περιορισμένη η έκταση του εγγράφου εργασίας, το χώρισα σε τρία μέρη. Το έγγραφο εργασίας ολόκληρο αποτελείται από τέσσερα μέρη, την εισαγωγή, την ανάλυση των προβλημάτων, τη βασική φιλοσοφία και τις αρχές, και τις επιμέρους μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Υποβάλλω 35 συγκεκριμένες προτάσεις στο έγγραφο που είναι αριθμισμένες. Το πρόβλημα, τα προβλήματα της κοινή ελευθερικής πολιτικής είναι γνωστά είναι η υπεραλίευση, η πτώση της οικονομικής ισχύω και της απασχόλησης, πλεονάζουσα αλλιευτική ικανότητα, κατασπατάληση των πόρων λόγω απόρριψης των παρεμπιπτών των αλλιευμάτων, συγκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Το τρίτο κομμάτι που είναι η βασική φιλοσοφία και οι αρχές μου είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει κατά την επίλυση των προβλημάτων να λάβουμε υπόψη μας το πρόβλημα της ανάγκης για συνοχή των μεταρρυθμίσεων. Τέλος, τα επιμέρους μεταρρυθμιστικά μέτρα, ε, λογικό είναι να είναι το εκτενέστερο κομμάτι αυτό. Ε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά να μην χάσουμε και τη φιλοδοξία μας. Στόχος της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ότι η βιομάζα των αποθεμάτων θα πρέπει να ε, αυξηθούν. Έχω τροποποιήσει λίγο την άποψη της Κομισιόν γιατί λέω ότι τα αποθέματα μέχρι το 2015 θα πρέπει να αυξηθούν ε, όσο είναι δυνατόν ε, α, στα όρια της μέγιστης απόδοσης, βιώσιμης απόδοσης. πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Κομισιόν θέλει να έχουμε πολυετή προγράμματα για το, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα προγράμματα το Συμβούλιο, δεν θέλει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε άλλους τρόπους. Προτείνω λοιπόν η αληθινισιμότητα να μειωθεί σε σχέση με τη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Στο βασικό κανονισμό θα πρέπει αυτό να είναι δεσμευτικό, και εδώ αναφέρομαι στην πρότασή μου υπαριθμών 3. Το 2015 ε, μπορεί να είναι εφικτό ως βιώσιμη απόδοση γίνεται αυτό γιατί όσο καλύ, ταχύτερα γίνεται η ανασύσταση τόσο περισσότερα λιεύματα θα έχουμε. Βέβαια θα περάσουμε από μεταβατική ε, φάση που θα πρέπει για ορισμένα αποθέματα να μειωθεί και δραστικά μάλιστα για ορισμένα είδη. Ιδιαίτερα ε, πληττόμενους θα πρέπει προσωρινά να τους ε, ενισχύσουμε γιατί δεν θα πρέπει λόγω των μεταβατικών μέτρων να κλείσει καμία αλληλευτική επιχείρηση. Αυτή η ιδέα μου είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν την αναφέρω στην πρότασή μου υπαριθμών 2. Αυτή την πρόταση θα πρέπει να τη συζητήσουμε πολύ και με τον συνάδελφο Καντέκ γιατί στο EFFF ε, θα βρούμε λύση. Ε, για την πέμπτη πρόταση, διαχείριση με βάση τη βιώσιμη απόδοση, αυτό θα γίνει μόνο όταν βελτιώσουμε τη συλλογή δεδομένων. Κάποια κράτη-μέλη δυστυχώς δεν συνεργάζονται όμως εδώ. Πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις και μέσα από αυστηρότερες κυρώσεις. Ε, τώρα, η απόρριψη, ε, η απόρριψη της επανάρριψης. Ε, αυτό έχει νόημα γιατί διότι ε, συνολικά θα ε, έχουμε περισσότερα αλλιεύματα. Δεύτερον, διότι τα αλλιεύματα θα ε, αφαιρούνται από την ποσόστοση, άρα θα έχουμε σωστή διαχείριση της ελίας. Τρίτον, έτσι η βάση των δεδομένων θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Θα πρέπει όμως να μπορεί να γίνει η πολιτική για την επανάρρηψη και να μην είναι και αντιπαραγωγική. Προτείνω λοιπόν την πρόταση 6, η απαγόρευση επανάρρηψης για όλα τα εμπορικά είδη θα πρέπει να εισαχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ε, δεν θα ισχύει για ψάρια που δεν μπορούν να τύχουν μεταποίησης. Βέβαια, δεν θέλουμε να γίνονται εκφορτώσεις ε, και μετά να ε, πετιόνται η έβδομη πρόταση, η απογόρευση επανάρρευσης θα πρέπει να γίνει ε, σταδιακά στην αλίευση και όχι με βάση τα είδη. Έτσι στα πολυετή προγράμματα για τα αλλιεύματα αυτά θα, πρέπει να, θα μπορούν να γίνουν οι προσαρμογές και των σχετικών κανόνων. Τέλος, ε, είναι σημαντικό να ισχύει μια γενικότερη ε, συνολική απόρριψη. Επίσης, θα πρέπει ε, να ε, όταν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της απόρριψης θα μπορεί να εφαρμόζεται σωστά από τους αλληλείς. Επίσης χρειάζονται πιλωτικά προγράμματα ούτως ώστε κάποιες επιλεκτικές σωστές πρακτικές να διαδοθούν και να διερευνηθούν και καινούργιες τεχνικές και τεχνολογίες. Πρόταση 9. Στα, ε, όποιος ψαρεύει ε, ηχθίδια θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο σε σχέση με την ποσόστοση. Ίσως αυτό ε, δεν ακούγεται πολύ ε, σωστό και ότι προσανατολίζεται κατά των αλλιέων. Όμως ε, ουσιαστικά η πρόταση σημαίνει ότι η συνολική ποσόστοση μπορεί ελαφρά να αυξηθεί και εκείνος που αποφεύγει τα, να ψαρεύει ε, ηχθίδια θα αμείβεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε τα παρεπιπτόντα αλλιεύματα να τα μειώσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι η μείωση των παρεπιπτόντων ε, θα πρέπει να γίνεται και να θεωρείται πιο σημαντική από την απόρριψη. Ε, τώρα, ε, με βάση την Ορβηγία η επόμενη πρόταση μπορούμε να ε, έχουμε ένα κίνητρο έτσι, 11. Η απαγόρευση της απόρριψης είναι αντιπαραγωγική και γι' αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις για παράδειγμα ως μέρος της μεταρρύθμισης αυτής ή μετά μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Είναι σημαντικό όμως η απαγόρευση των απορρίψεων να ισχύει και μετά για επιμέρους ήδη, σε μεμονωμένους τρόπους αλληλείας ε, να προβλέπονται εξαιρέσει, όχι αντίστροφα. Στο έγγραφο εργασία μου υποβάλλω και κάποιε προτάσει, ε, πρόταση 12, 14 και 16, για το πώς μπορούμε το πρόβλημα της κατανομής των ποσοστώσεων με το αξί των ε, κρατών μελών να το λύσουμε. Αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να είναι το έναυσμα για τη συζήτηση. Θα πρέπει από κοινού με το Συμβούλιο να επιχειρήσουμε να βρούμε ένα σωστό και δίκαιο σύστημα. Θέλω να τονίσω ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταλάβουν ότι εμείς ε, λόγω εθνικών εγωισμών κάνουμε απορρίψεις. Είμαι βέβαιη ότι στο τέλος θα βρεθεί λύση. Τώρα πάμε στο, σημείο, στο μέρος 3 του εγγράφου εργασίας και στο μεγάλο θέμα ε, των μεταφερόμενων αλληλευτικών εκχωρήσεων. Εδώ πρέπει να βρούμε καλές λύσεις, ε, έξυπνες. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για, για ένα θέμα που μέχρι τώρα δεν το έχουμε συζητήσει. Για τα πλεονεκτήματα των μεμονωμένων ατομικών ποσοστώσεων. Ατομικών λέω πολύ συνειδητά όχι ε, ατομικά μεταβιβάσιμων ε, ποσοστώσεων. Η τήρηση των ποσοστώσεων από το εκάστοτε κράτος μέλος θα μπορεί να ελέγχεται καλύτερα από ότι αν υπήρχε μια συνολική κρατική ποσόστοση. Σε τέτοιες περιπτώσεις το κράτος θα πρέπει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να ε, κλείνει ε, ζώνες ε, αλίας. Αυτό, πολλές αυτό πρέπει να γίνεται όμως στην πραγματικότητα. Επίσης, έχουμε το περίφημο Race for the Fish. Οι αλίες προσπαθούν να αυξήσουν τα αλληλεύματα... όσο γίνεται περισσότερα. Και κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε κακό καιρό, βγάζουν τα πλοία έξω. Στις ατομικές ποσοστώσεις όμως, ο αλίας από μόνος του μπορεί να αποφασίσει πότε θα αξιοποιήσει την ποσόστοσή του με τον καλύτερο τρόπο. Ε, θα, ε, ε, ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας επάνω εδώ και τη γνώμη της Κομισιόν βέβαια, γιατί μέχρι τώρα αυτό το θέμα δεν το έχουμε σχεδόν καθόλου συζητήσει. Ε, τώρα, Ε, όταν υπάρχει ε, υπερβάλλον ελιευτικό δυναμικό, ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, επαναπροσδιορισμού της. Η πλεονάζουσα ελιευτική ικανότητα θα πρέπει να μην υπολογίζεται με βάση τον όγκο και την ισχύ του κινητήρα των ε, σκαφών. Η αλλιευτική ικανότητα όμως εξαρτάται επίσης και από τα ε, σκάφη και τον εξοπλισμό τους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, την αξιολόγηση αυτών. Όπου υπάρχει πλεονάζουσα αλλιευτική ικανότητα θα πρέπει να υπάρχει και μια υποχρέωση σε πολλές περιπτώσεις ε, ένα μέσον θα ήταν ε, ένα σύστημα ε, TFC για τους αλληλείς. Δηλαδή, αν αποδεικνύει το κράτος μέλος ότι την μείωση της ικανότητας μπορεί να την έχει χωρίς ε, ε, τα τάκα, ε, θα, πρέπει να μπορεί να την κάνει. Εδώ παραπέμπω στην πρόταση 19. Είμαι έτοιμη να παρεκκλίνω από ένα υποχρεωτικό σύστημα τάκα, αλλά με την προϋπόθεση μόνο ότι θα πρέπει οι ικανότητες να αξιολογηθούν και όταν αυτές παρουσιάζουν πρόβλημα να μειώνονται όντως. Οπουδήποτε ε, εισάγονται τάκ θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το σύστημα θα πρέπει να διαμορφώνεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις να αποφεύγονται. Αυτή την ιδέα την παρουσιάζω στην πρόταση 21. Σημαντικό είναι ότι κατά τη διαμόρφωση ενός συστήματος TFC ε, οι αλληλείς, ιδιαίτερα οι μικροί αλληλείς, να συμμετέχουν και αυτοί. Αυτό είναι ο βασικός μου προσανατολισμός. Ε, χαίρομαι που θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή και πιστεύω ότι θα συζητήσω με επισωστής βάσεως. Τέλος, το 4-4, η περιφερειοποίηση. Εδώ ε, τα πολιετή προγράμματα είναι το βασικό. Για να επιτευχθούν ε, οι στόχοι μας ε, προϋποτίθεται βελτιωμένη ε, συμμετοχή όσων συμμετέχουν στην χάραξη αυτών των προγραμμάτων. Πρόταση 23. Οι νομοθέτες εδώ δεν θα πρέπει να κάνουν μόνο δηλώσεις, αλλά να προβλέπουν ότι οι εμπλεκόμενοι κατά την επεξεργασία μιας πρότασης της Κομισιόν για να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις θα πρέπει τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, τα ΡΑΚ, να παίζουν σημαντικό ρόλο, πρόταση 24. Προϋπόθεση όμως είναι η σύνθεσή τους να γίνει πιο αντιπροσωπευτική και οι εργοδότες, οι καταναλωτές ε, και τα περιβαλλοντικά συμφέροντα να ενισχυθούν. Και η επιστημονική διαβούλευση των ΡΑΚ, των γνωμοδοτικών συμβουλίων, πρέπει να βελτιωθεί. Πρόταση 25. Τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται κατά την ε, έγκριση των εθνικών μέτρων να συμμετέχουν. Αυτή η συμμετοχή ε, μπορεί να συντονίζεται από την Κομισιόν και η πρόταση 26, η στόχοι που ορίζει η Κομισιόν θα πρέπει να ε, πραγματοποιούνται, να υλοποιούνται. Ε, δεν ξέρω εδώ αν τα προτινόμενα όργανα ελέγχου επαρκούν. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόταση 27. Αν πούμε ότι με την έγκριση της μεταρρυθμιστικής δέσμης θα πρέπει να ε, ολοκληρώνεται ο έλεγχος ε, θα πρέπει ε, να μπορούμε κάποιους ευρωπαϊκούς κανόνες να τους ε, καταργούμε αν δεν είναι αναγκαίοι. Θα πρέπει όμως να γίνονται όλοι οι διαχειριστικοί έλεγχοι. Αυτές είναι οι σκέψεις από αυτού του θέματος. Ως Επιτροπή όμως θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε, να αναθέσουμε στην νομική υπηρεσία να εξετάσει αν και πώς ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην περιφερειοποίηση. Το έγγραφο εργασίας έχει και ένα πρόσθετο κεφάλαιο για τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Επειδή η κατάσταση κατάσταση εδώ διαφέρει από εκείνη της υπόλοιπης Ευρώπης. Τα αποθέματα τα ηχθείων σε μεγάλο βαθμό αλλιεύονται παρακτίως. Υπάρχουν ε, λίγα αποθέματα τα οποία αλλιεύονται ταυτόχρονα από πολλές χώρες. Και η δομή του στόλου διαφέρει από εκείνον του Ατλαντικού και της Βόρειας Ευρώπης ε, γιατί είναι ε, μικρότερης κλίμακας. Η μεταρρυθμιστική πρόταση εδώ θα πρέπει να βελτιωθεί πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέσα, ε, μέτρα που θα συμπληρωθούν για να λάβουν υπόψη τον εύξηνο πόντο και τη Μεσόγειο. Υποχρέωση, για παράδειγμα, ε, ενό δικτύου ε, κλειστών περιοχών άβατων περιοχών. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε ειδικά για τη Μεσόγειο. Ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα για να ε, διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις και ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Η το Η ιδέα που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν είναι η δημιουργία ενός Συμβουλίου για την υδατοκαλλιέργεια και η δημιουργία μη υποχρεωτικών κατευθυντηρίων γραμμών για κοινέ προτεραιότητε και στόχου. Αυτό είναι προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι προτάσει αυτέ δεν επαρκούν για να ε, ε, δώσουν την απαραίτητη δυναμική στον τομέα αυτόν που έχει στασιμότητα. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε πιο ανταγωνιστικό. Για να επιτύχουμε τους στόχους θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι προβλέπει, από ό,τι να αλλάξουμε το βασικό κανονισμό. Όμως ε, οι ακόλουθοι στόχοι μπορούν να ε, συμπεριληφθούν στο βασικό κανονισμό, ούτω ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την περαιτέρω βελτίωση. Πρόταση 30, θέσπιση πιο αυστηρών ε, ποιοτικών κριτηρίων, ε, διαφανών και γενικών, σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια, που θα εξασφαλίζονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία θα διασφαλίζουν τις οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας. Πρόταση 31 Εκεί λέω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες σχετικά με την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και 32 πρέπει να υπάρξουν ε, κριτήρια επισήμανσης για υψηλής ποιότητας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και για βιολογική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας πιο συμβατή με το περιβάλλον. Πρόταση 33 ε, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας θα παράγονται σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές ποιοτικέ προδιαγραφές, όπως οικολογικές προδιαγραφές και προδιαγραφές για την ευζοία των ζώων. Πρόταση 34, ε, διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας για βιώσιμη από περιβαλλοντικής πλευράς υδατοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόταση 35. Χρειαζόμαστε μία πρωτοβουλία για την ε, μείωση της γραφειοκρατίας. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι η μείωση της γραφειοκρατίας θα πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε το σύνορα. Ε, προσβλέπω με χαρά στη συμβολή σας και στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρόντουστ. Θα ξεκινήσουμε τώρα δίνοντας το λόγο σε όσους το επιθυμούν. Κύριε Στίβενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ρόντουστ ανέλαβε τη δυσκολότερη έκθεση στην ιστορία της Επιτροπής μας και είναι σαν μουσική ακούγεται στα αυτιά μου τώρα που την άκουσα να την παρουσιάζει, την έχω φυσικά διαβάσει, αλλά ήταν καταπληκτικές οι εισαγωγικές της ε, παρατηρήσεις. Συμφωνώ σχεδόν ε, με όλα τα σημεία που συμπεριέλαβε. Πρώτον, Συμφωνώ να επιλέξουμε μέχρι το 2015 την μέγιστη βιώσιμη απόδοση που βασίζεται στην εθνισμότητα των ψαριών. Ε, νομίζω ότι ούτως ή, άλλως, ο, ούτως ή άλλως συμφωνούσαμε, αλλά δεν ε, μπορούσαμε να πετύχουμε την άλλη μέγιστη βιώσιμη απόδοση που βασίζεται στη βιομάζα, διότι ήταν πάρα πολύ στενό το χρονοδιάγραμμα. Τη δεύτερη όμως μπορούμε να την επιτύχουμε. Τώρα υπάρχει και το θέμα της μεικτής αλληλείας ε, που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Λέτε ότι φέτος θα εισαγάγουμε παραδείγματος χάρη για τις απορρίψεις μπακαλιάρου μία απαγόρευση και του χρόνου το ίδιο για τον ε, εγκλεφίνο. Ε, ε, αλλά συγγνώμη, μιλάμε για μεικτή αλία, άρα αλλιεύονται ε, πολλά είδη και νομίζω ότι γι' αυτό αιτιολογείται η προσέγγιση σας και συμφωνώ. Επίσης, συμπεριλάβατε ε, μερικές πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλίες καθημερινά, το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω. Αν έχετε απομακρυνθεί από το λιμένα εκατοντάδες ε, χιλιάδες μίλια και έχετε πολύ περιορισμένο ε, αριθμό ε, ημερών αλίας βάσει του περιορισμού των αλλιευτικών δυνατοτήτων και αλλιεύσετε μικρό ψάρι, και επειδή ισχύει αυτή η απαγόρευση θα πρέπει να τα απορρίψετε και πάλι αυτά τα μικρά ψάρια πριν φτάσετε στο ε, λιμάνι, να θα έχουν βρωμίσει στο μεταξύ. Να τα πάμε στη χωματερή καλύτερα. Ε, πρέπει ε, στα μέτρα που προτείνουμε να έχουμε κατά νου την πραγματικότητα, τις πρακτικές δυσκολίες καθημερινές ε, για τους ψαράδες. Επίσης υπάρχει το θέμα της εκφόρτωσης των ηχθείων που δεν έχουν φτάσει σε όριμη ηλικία και συμφωνώ με την πρότασή σας διότι με τη νέα πρόταση θα μειωθούν τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα και έτσι θα αποκτήσει ένα νόημα η όλη έννοια της απαγόρευσης των απορρίψεων. Συζητήσαμε και με τους το θέμα αυτό θεωρούν ότι ε, έχουμε περίπου 50% απορρίψεων στον κλάδο τους, στον κλάδο της αλίας και επανέρχομαι σε αυτά που σας έλεγα με τα βρωμερά ψάρια ε, και το, το παράλογο του να πρέπει να εκφορτωθούν αυτά. Ε, για τα για τις ε, μεταβιβάσιμες ε, αλλιευτικές ε, παραχωρήσεις. Νομίζω ότι με αυτή την ρήτρα διασφάλισης είναι η σωστή οδός, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. 50 χρόνια νομίζω θα ήταν πλημελής λύση. 7-8 χρόνια και όχι 15 θα πρέπει να προτείνουμε για τις μεταβιβάσιμες αυτές παραχωρήσεις. Επίσης χρειαζόμαστε αυστηρές εγγυήσεις για τα ψάρια. και αυτό θα καλύπτεται από την μη υποχρεωτική προσέγγιση που ε, ε, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας δούμε και το επιτυχημένο δανεικό πείραμα, δηλαδή μικροί ψαράδε δίνονται να αγοράσουν βιβάσιμη ποσόστοση από ε, τους μεγάλους αλληλεί, αλλά το αντίστροφο δεν είναι δυνατόν. Είδου λοιπόν μια δικλίδα ασφαλεία, Τέτοιε χρειαζόμαστε. Ε, τώρα, Ε, για, ε, είμαι πεπισμένος ότι μόνο 6,7 δις προβλέπονται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον ε, τομέα της αλίας και θα πρότεινα να εξετάσουμε την επανεσαγωγή κάποιων επιδοτήσεων διότι ως προς τον εξυγχρονισμό του στόλου ε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε και άλλες δυνατότητες πέρα δηλαδή από τον εξυγχρονισμό του στόλου μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν τα σκάφη ε, θα πρέπει να είναι εμπορικά, και, εμπορικά κερδοφόρα η επιχείρηση, αλλιώς ε, δεν είναι βιώσιμη. Και εάν χρειάζεται κάποιος μία επιδότηση για να είναι κερδοφόρος, καταλαβαίνετε ότι θα κλείσει αν δεν πάρει αυτή την επιδότηση και έτσι θα επέλθει αυτή η μείωση του στόλου που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία έχουμε συμφωνήσει και εμείς. Οπότε, εάν ε, επιλέξουμε αυτήν την άγουσα της ε, επιδότησης ε, του εξυγχρονισμού του στόλου ή του εξοπλισμού, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι με τον εξχωνισμό των κινητήρων ε, των ε, σκαφών θα μειωθούν οι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, τώρα που είναι πολύ ακριβά τα καύσιμα, θα είναι πιο αποτελεσματικό το σκάφο. Με καλύτερο κινητήρα θα λιευθούν όμω και περισσότερα ψάρια και δεν είναι ο στόχο μα. Οπότε θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Εξάλλου το αναφέρει και η Επιτροπή στο έγγραφό Πιστεύω ότι ε, το σημαντικό σε σχέση με το στόλο μικρή κλίμακας και όχι βιομηχανικής, όπως λέγαμε και έχουμε επανειλημμένα αναφέρει στην Επιτροπή μας, ε, πρέπει να τονιστεί όντως, ε, αλλά και πάλι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να αποφασίσουν για το τι κάνουμε τι στρατε τους μέσα στα όρια των 12 μιλιών. Δεν νομίζω ότι ε, μιλούσατε ουσιαστικά για τις οχθοκαλλιέργειες, όταν μιλούσατε για τη μείωση τη γραφειοκρατίας, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε μείωση τη γραφειοκρατίας ε, σε σχέση με αυτή τη μικροδιαχείριση που επιχειρείται από πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, θα έπρεπε να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Το ίδιο ισχύει και για την περιφερειοποίηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εμπλακούν όλα τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη και όπω λέτε στην έκθεσή σα. Ε, κυρία Ρόντουστ, θα πρέπει να αποσκοπούμε και στην ενίσχυση των υφιστάμενων περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων, γιατί έχουν σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά χρειάζονται ε, περισσότερη πυγμή, μεγαλύτερη ισχύ. Ε, το ίδιο νομίζω ισχύει και για την ηχθειοκαλλιέργεια ε, όπως έχουμε το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τα βενθικά είδη ή για τη Βόρειο Θάλασσα, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την ηχθειοκαλλιέργεια. Χρειαζόμαστε ξεχωριστές ποσοστώσεις και ξεχωριστές το προσωπικό, διότι είμαστε αυτόνομοι μόνο σε ποσοστό 40%. Δηλαδή, εισάγουμε 60% των ψαριών από τρίτε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διοικητεύσουμε του πόρου μα στην ε, περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου τη ηχθειοκαλλιέργεια. Κάνοντα αυτό, θα μειώσουμε και την γραφειοκρατία και έτσι θα έχουμε ένα ε, γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ηχθειοκαλλιέργεια που θα είναι ουσιαστικό. Ε, είναι εξαιρετική η έκθεσή σας και σας συγχαίρω. Ευχαριστώ. Κυρία Λεβάν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ρόντους για όλη τη δουλειά που έκανε. Πραγματικά είναι πολύ θετικό το έργο σας και το, να διαβάζουμε το έγγραφο εργασία σας ε, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία που αναφέρετε. σα συγχαίρουμε λοιπόν για την καλή δουλειά. Θα ήθελα να δούμε όλα τα κυρία σημεία Καταρχήν, να πω ότι υποστηρίζουμε την προσέγγιση για το FMSY με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για την θυσιμότητα των ψαριών και με το στόχο να πετύχουμε το BMSY, δηλαδή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τη βιομάζα και επίση τη δυνατότητα να έχουμε ε, στο βασικό κανονισμό εισαγωγή κανόνων ε, για τον έλεγχο τη ελίευση τη οδειά, καθώ τα σχέδια διαχείριση ε, δεν παρέχουν την απαρκή ασφάλεια. και δεν μας επιτρέπουν να προοδεύσουμε όπως θέλουμε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ βασικό που πρέπει να έχουμε στο βασικό κανονισμό σε ό,τι αφορά τώρα τα περιπτώτα αλλιεύματα. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση ε, όχι ανά είδος, αλλά ε, ανά αλία και αναφέρατε τα εμπορικά είδη, αλλά πιστεύουμε ότι όλα τα είδη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα μη εμπορικά αλλά βέβαια να αποκλείσουμε όσο μπορούν να επιβιώσουν. Και αυτό που νομίζω ότι λείπει και στην πρόταση της Κομισιόν. Και το ανέφερε εδώ κύριο, το έδωσε έμφαση στη μείωση των περιπτωτών ελευμάτων. Νομίζω ότι όλα τα κρατημέλη θα πρέπει να υποχρεούνται επίση να προτείνουν ένα σχέδιο για την μείωση των περιπτώτων ελευμάτων. Δεν θα πρέπει να είναι σε ακούσια βάση δηλαδή. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε νέα αγορά για τα μη εμπορικά είδη και τώρα θα τα καταστήσουμε ήδη στόχους και να μην ε, δίνουμε χρήματα για ε, την μεταποίηση αυτών ε, των αλλιευμάτων. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια πρόταση βάση ε, ε, Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα μειώσουμε τα παραλιεύματα. Γιατί αν απλώ λέμε ότι πρέπει όλα να εκφορτώνονται, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα προσπαθήσουν οι Έλληνες να αποφύγουν τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα και αυτό είναι ο στόχος όλων αυτών. Να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα σε σχέση και με τις ποσοστώσεις ε, των παραλιευμάτων. Διστάζω λοιπόν κάπως ε, για την πρότασή σας ε, στο σημείο 16, δηλαδή να μεταφέρουμε τις ποσοστώσεις παραλιευμάτων από το ένα έτος στο άλλο. Δεν θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα των κανονικών υπολογισμών των τάξ αλλά αν έχετε μία ποσόστοση για τα παραλίευματα, ίσως δεν θα έπρεπε να είναι μία πρόσθετη ποσόστοση, ούτε θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να εμπορευόμαστε. Ε, για την ε, υπερβολική ελευτική ικανότητα. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Κάτι που δεν έχει συζητηθεί ε, είναι τα ανώτατα όρια της ικανότητας. Τώρα έχουμε τέτοια όρια από το 2003 και είναι πολύ πιο πάνω από ε, το ανώτατο ε, που έχουν τα κράτη-μέλη και είναι κάπως στον αέρα αυτό το ανώτατο. Έτσι λοιπόν πρέπει να ε, αφαιρέσουμε τον αέρα, ε, για να το πω έτσι, και πρέπει να δούμε πόση ικανότητα υπάρχει. Υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Ρόντουστ ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση αναλύευμα για την πραγματική ελευτική ικανότητα και πόση πλεονάζουσα ελευτική ικανότητα υπάρχει. Νομίζω ότι αυτή είναι καλή ιδέα αλλά Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο της αλληλευτικής ικανότητας γιατί αν ορισμένα κράτη-μέλη επιλέξουν ε, να μην ε, συμπεριλάβουν ε, τα TFCs, δηλαδή τις μεταβάσιμες αλληλευτικές παρακολουθήσεις, χρειαζόμαστε εργαλεία για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι στη Σουηδία έχουμε εισαγάγει ITQs στα πελαγικά αλλιεύματα και το 50% ε, της ε, ικανότητας ε, αφαιρέθηκε στη Σουηδία, αλλά η ονομαστική ικανότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Έτσι λοιπόν κάθονται στις αποβάθρες αυτά τα σκάφη και αν υπάρχουν πρόσθετες ελευτικές ικανότητες για αυτούς τους ελείς, τότε μπορούν με τα δικά τους χρήματα να παροπλήσουν αυτά τα σκάφη και να φτιάξουν ένα νέο σκάφος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την ικανότητα, μείωση της ικανότητας σε κιλο... κιλοβάτ. Διαφορετικά υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν νέα σκάφη στο μέλλον και για τον Εύξηνο Ποτό και για τη Μεσόγειο. Για να τελειώσω, είμαστε πολύ διστακτικοί, δεν μας αρέσει να δημιουργήσουμε δύο διαφορετικά πρότυπα για τον Ευξηνό Πόντο και τη Μεσόγειο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ίδια για όλους ε, σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, ε, την πολιτική, τα μέτρα διατήρησης. Ε, πρέπει όλα αυτά να είναι τα ίδια γιατί διαφορετικά θα δημιουργήσουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων στην Αλία και δεν θέλουμε να το δούμε αυτό. Και η πρόταση για τι προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχές. Ε, το υποστηρίζουμε, αλλά θα πρέπει να ισχύει για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Μεσόγειο, για τον Ευξηνοπόντο. Πόντο. Και νομίζω ότι εδώ θα κλείσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή. Χάτκον. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μετά από την κυρία Λόβιν, είμαστε συνάδελφοι στην ομάδα, θα προσθέσω ότι υπάρχει ένα σημείο επί το οποίο μάλλον ε, καταρχάς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, γιατί δεν χρειαζόμαστε προσέγγιση δύο ταχυτήτων, πολλαπλών ταχυτήτων χρειαζόμαστε σε αντίθεση με την κοινή προσέγγιση του παρελθόντος, σε αντίθεση με την κεντρική κεντροποιημένη προσέγγιση με μία λύση ενιαία για όλους που έχουμε ήδη υιοθετήσει στο παρελθόν. Πιστεύω πραγματικά ότι πολλές από τις δυσκολίες που αναγνωρίζουμε όλοι και σίγουρα όλοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αμέσως απότοκες ε, αυτού του γεγονότος. Ε, δηλαδή ότι θέλουμε να θεωρήσουμε κάποιες περιοχές ε, και κάποια είδη ψαριών ως ταυτόσημα ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές λόγω κλίματος, λόγω ιδιαιτεροτήτων της θαλάσσιας περιοχής και άρα θα πρέπει ό,τι όποια προσπάθεια κάνουμε για τη διατήρηση του αποθέματος να προσαρμόζεται στην κάθε περιοχή και στο κάθε είδος, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, κυρία Ρόντες, τούτου λεχθέντος, ε, δεν ε, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να διαβάσουμε μέσα από τις γραμμές ε, και να πούμε εντάξει η υπεραλίευση είναι κάτι το αρνητικό και πρέπει να το καταπολεμήσουμε, η απόρρεψη είναι σκάνδαλο και αυτό πρέπει να το καταργήσουμε, η πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα το ίδιο, πρέπει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση για να την αντιμετωπίσουμε και το καθεξής και σίγουρα εγώ θα ταχθώ υπέρ της αποκεντρωμένης προσέγγισης, αλλά θα άρχιζα από αυτό. Από αυτό θα άρχιζα, από την αποκεντροποίηση και στη συνέχεια θα άρχισα να αντιμετωπίζω αυτά τα βασικά προβλήματα του κλάδου της αλίας, διότι όπως προείπα, η ε, βασικέ διαφορέ ανάμεσα στι θαλάσσιε περιοχέ και στα είδη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το δέοντα τρόπο, εάν θέλουμε να σημειώσουμε επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα που τώρα ξεκινάμε ε, από την εμπειρία που έχω εγώ από την κοινή αλληλευτική πολιτική, συναγάω το εξή συμπέρασμα, ότι αν θα επιθυμούμε ε, να αναβαθμίσουμε τη διαχείριση των αλλιευμάτων στο μέλλον, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ και όχι να κάνουμε μία ε, εκβάθρον ε, μεταρρύθμιση του συστήματος. Τι σημαίνει αυτό. Η αλληλευτική τα αλλιευτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ισχύ, ούτω ώστε ε, με τις αρμοδιότητες τους να μπορέσουν να διαχειριστούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τι ε, θαλάσσιες περιοχές και τα είδη που αλλιεύουν. Ε, Επίση, θα πρέπει να δούμε πώ ακριβώ θα συντονιστεί η αλληλεία γειτονικών χωρών. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε φυσικά τα διασυνοριακά ζητήματα για κάποια μεταναστευτικά είδη. Ε, όπως λέει και η ΆΙΚΑΤΕ για τις ε, θαλάσσιες ε, λεκάνες υπάρχουν πολλοί λογικά επιστημονικά δεδομένα και υπάρχουν κάποια προβλήματα που μπορούμε να ρυθμίσουμε κεντρικά και άλλα όχι. Όσοι έχουν δικαιώματα στη Βαλτική, παραδείγματο χάρη, δεν είναι παράλογο να καταβάλουν σκληρές προσπάθειες ούτως ώστε να είναι βιώσιμη η αλληλεία τους για το μέλλον. Αν κάποια στιγμή ε, στο μέλλον, όπως τώρα προτείνεται για την κινητική πολιτική, θέλουμε να εξασφαλίσουμε κοινή πρόσβαση στους αλληλευτικούς πόρους. Ε, δεν τους ενθαρρύνουμε έτσι αυτούς που έχουν δικαιώματα αυτή τη στιγμή στη Βαλτική ε, να κάνουν τι προσπάθειες για το δικό τους μακρόπνο όφελος. Ε, ως προς τις απορρίψεις. Ε, πολλά από αυτά που λέγονται για τις ε, απορρίψεις εδώ και αλλού ε, είναι ορθά, είναι σκάνδαλο, είναι απευκταίο τα νεαρά ηχθίδια να παραλιεύονται και στη συνέχεια να απορρίπτονται και να θέτουμε σε κίνδυνο τα αποθέματα. Μην ξεχνάτε όμως πως κάποιοι από τους ισχύοντους κανονισμούς της τωρινής κοινής αλληλευτικής πολιτικής οδηγούν άμεσα σε απόρριψη ε, μεγάλων ψαριών, όριμων ε, ψαριών, ε, διότι ψαρεύουν εγκλεφίνο και έχει μπακαλιάρο δίπλα. Ο μπακαλιάρος είναι μεγαλύτερος, είναι δύσκολο ο ψαράς να μην πιάσει και τον μπακαλιάρο. Οπότε όταν μιλάτε για τις απορρίψεις, μιλάτε μόνο για ψάρια που δεν έχουν εμπορική αξία ή που είναι πολύ μικρής ηλικίας. Δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα και θα ήταν δύσκολο, ε, λάθος ε, να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, δηλαδή άχρηστα ψάρια να εκφορτώνονται, ε, γιατί βάζει το, το ε, στην ξηρά, ενώ τώρα τι, εκφορτώνονται, απορρίπτονται στη θάλασσα. Το ίδιο είναι. Τι σημαίνει αυτό, περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερες εργασίες, ε, καλύτερες επιστημονικές συμβουλές, ε, ακρίβεια, καλύτερες επιστημονικές προβλέψεις. Αυτό είναι που αντίθετα χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο και να βρούμε μια ε, ποσοστώσεις που, πώς να το πω, θα είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα για να μην οδηγούν σε απόρριψη εδόδημων και με μεγάλη εμπορική αξία ειδών ψαριών. Για τις ε, μεταβάσιμες ποσοστώσεις αυτή τη στιγμή ε, μάλλον να το πάλι αλλιώς, ε, δίκαιο έχει η κυρία στο που ανέφερε το θέμα της ατομικής ευθύνης. Νομίζω ότι βοηθάει αυτή η έννοια, η σκοτία από την οποία προέρχομαι, φέρει μια μεμονωμένη ευθύνη, διότι έχουμε την ποσόστοση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ανακατανέμεται προ την Σκοτία ε, και άλλε περιοχέ ε, και στη συνέχεια γίνεται κατανομή ανασκάφο ε, σε διάφορες δηλαδή αλληλευτικές επιχειρήσεις, ε, κατανοήμονται οι ποσοστώσεις και αυτές ε, ε, οι εκμεταλλεύσεις είναι υπεύθυνε για την ποσόστοσή του για τη διαχείρισή της και άρα καλούνται να πάρουν τις σωστές αποφάσεις το ώστε μακροπρόθεσμα να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Όμως ανακύπτουν δυσκολίες και δεν προκύπτει άμεσα πώς με την βιώσιμη διατήρηση του αποθέματο θα έχουν κάποιο κέρδος στο μέλλον. Σχετικά τώρα με ε, τις μεταβιβάσιμες ε, αλλιευτικές ε, παραχωρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε αυτή την πρόταση και μας είπε ότι να η απλή και αποτελεσματική λύση για την πλεονάζουσα ε, αλλιευτική ικανότητα. Όπω σωστά υπέδειξε η κυρία Ρόντουστ, θα πρέπει να κάνουμε πριν αποφασίσουμε την δέουσα αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση, μάλλον να εντοπίσουμε πού ακριβώ εντοπίζεται αυτή η πλεονάωσα αλλιευτική ικανότητα. Αυθαίρετα και ε, από το κέντρο, από τις Βρυξέλλες, ε, θα αποφασίσουμε ότι όλοι έχουν πρόβλημα πλεονάζουσας αλλιευτική ικανότητα. Υπάρχουν κάποιοι που το έχουν ρυθμίσει το πρόβλημά σε προηγούμενε τη κοινή κοινή αλληλευτικής πολιτικής εισηγήτρια ε, σωστά ανέφερε ότι ε, υπάρχουν υπέρ και κατά με το νέο σύστημα ακόμη και για αυτούς που έχουν ήδη ρυθμίσει το θέμα της ε, πλεονάζουσας ικανότητας και θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή να αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Η Δανία είναι το καλύτερο παράδειγμα βάσει και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εφαρμόσει, υποτίθεται, ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα. Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε μέσω κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εθνική πολιτική έγινε. Η Δανία ε, σχεδίασε ένα σύστημα ειδικά προσαρμοσμένο στην κατάσταση που επικρατεί στην Δανία. Για, για ποιο λόγο ε, λοιπόν να επέμβουν οι Βρυξέλλες σε σχέση με την μεταβιβασιμότητα των αλλιευτικών παραχωρήσεων. Νομίζω ότι τα κατά μακροπρόθεσμα θα είναι μοιραία για τον κλάδο και η κεντρική αντιμετώπιση των ζητημάτων για μια εμπορική δραστηριότητα που έχει τόσο κέρια σημασία για νησιώτικες και παράκτιες περιοχές ε, και ε, περιοχές όπως η Σκοτία και θα είναι μόνο θέμα χρόνου δυστυχώς προτού να καταστραφεί, αυτή, να καταστραφεί αυτός ε, ε, ο κλάδος ε, λόγω της υποχρεωτικής και αυθαίρετης, ξαναλέω, προσέγγισης που θα προέρχεται από τις Βρυξέλλες, καταστρέφοντας έτσι όλες τις παράκτες περιοχές. Σε σχέση με τη συμπερίληψη της ηχθειοκαλλιέργειας ή όχι, εκνευρίστηκα, θα το πω έτσι ήπια, η κοινή αλλιευτική πολιτική είχε τόσο κακές επιδόσεις στο παρελθόν που ελπίζω ε, να φτάσουμε επιτέλους στο σημείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθούμε τα κράτη-μέλη να αναβαθμίσουν αν θέλουν τον τομέα της ηχθειοκαλλιέργειας αλλά σε καμία περίπτωση σε κάθε λεπτομέρεια να τον ρυθμίσουν με νέους κανονισμούς και πάλι εδώ οι τοπικές και εθνικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση να ε, ρυθμίσουν την ηχθειοκαλλιέργεια. Ναι, μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, εντάξει, ποιος θα αντιτάξει σε αυτό κάποιο επιχείρημα, αλλά και πάλι εδώ... Ε, ας δούμε και ε, Ας δούμε ποια γραφειοκρατία απορρέει από την ίδια την αντίληψη ότι πρόκειται για κοινό πόρο. Όλοι αυτοί οι η πόροι δηλαδή της Ένωσης θεωρούνται ως κοινό πόρος και με υποχρεωτικό και αυθαίρετο τρόπο εμείς προσπαθούμε να τον ρυθμίσουμε και πιστεύω ότι αν δεν προσέξουμε θα είμαστε αντιπαραγωγικοί αντί να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κύριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως ε, και προλαλήσαντες, ε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι σε αυτό το έγγραφο θέτει κάποιες ε, πολύ ενδιαφέρουσες και καινοτόμες προτάσεις που συμπληρώνουν τις προτάσεις της Κομισιόν. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτες και μας βοηθούν. Και επίσης συνειδητοποιώ ότι είχαμε ένα-δυο Σκοτσέζους που πήραν το λόγο για ένα Βρετανό <laughs> ένα Γερμανό και κάποιο από τη Σουηδία θέλουν να τοποθετηθούν για κάποια από τι χώρε τη Μεσογείου για να δούμε αν συμφωνούν με την έκθεση αυτή και έχουν παρόμοιο ενθουσιασμό. Τώρα, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, μου αρέσει η πρόταση της εισηγήτρια. Δεν είμαι σίγουρος ε, για το να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το BMSY, το συντομότερο δυνατόν. Είναι κάπως να η διατύπωση αυτή και ελπίζω ε, να μπορέσουμε ε, να βρούμε έναν τρόπο να δεσμεύσουμε την Κομισιόν σε κάποιες δεσμεύσεις. Τώρα, για την απαγόρευση ε, των παραλιευμάτων. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς μια απαγόρευση των παραλιευμάτων όλων των ψαριών, όχι μόνο των εμπορικών ειδών, αλλά υποστηρίζω ένθερμα την ιδέα να το δούμε ένα λίευμα. Και εδώ έχουμε και ένα πολιτικό ε, επιχείρημα. Είπε η συγκεκριτρία ότι οι πολίτες μας δεν θα καταλάβουν αν ε, εμείς επιτρέψουμε ε, να συνεχίζονται τα παρελεύματα λόγω εθνικής, εθνικού εγωισμού. Όμως, κοιτάξτε, να έρθει και τη σκοτή και να πει εντάξει, όλοι θέλουμε την απαγόρευση των περιλημμάτων, αλλά δεν είναι ακόμα εφικτό. Αλλά εγώ αν πάω στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ, να μιλήσω εκεί Στου ανθρώπου ανθρώπους, όπου οι άνθρωποι τρώνε τα ψάρια, δεν τα αλλιεύουν και ζουν ε, σε μεγαλύτερα νούμερα, γιατί έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό, θα πούνε δεν μπορούμε να ανεχθούμε τα παρελεύματα, είναι ανήθικο, είναι κάτι κακό και είναι πολύ διαφορετική στάση. Έτσι λοιπόν, εδώ ίσως ε, στην Επιτροπή ε, να εκπροσωπείται ε, η άλλη, η προηγούμενη άποψη και όχι αυτή τη ε, πλειοψηφία όσο καταναλώνουν ψάρια. Τώρα για τι μεβέ αλληλευτικές παραχωρήσεις. Ήταν ε, κάτι αμφίσιμο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, και φυσικά υπάρχουν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ε, εγώ κατέθεσα μια τροπολογία η οποία ε, αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον εννέα διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ένα κράτος μέλος καθορίζει τις δικές του TFC και θα μπορούσε να συμπεριλάβει περιορισμούς για να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις ανησυχίες που έχουν αναφερθεί πολλάκις. Λόγου χάρη, τα κράτη-μέλη μπορούν να εισαγάγουν μια ε, TFC, μια τέτοια παραχώρηση που να περιορίζει την μεταβίβαση των ε, λευτικών περιχωρησιών μεταξύ τμήματων του στόλου, παραδείγματο χάρη μεταξύ μικρού και μεγάλου στόλου πελαγικών ειδών, ευηθοβίων ειδών. Θα μπορούσαμε να έχουμε ωρία για να προστατεύουμε γεωγραφικέ ε, περιοχέ όπω γίνεται στην Ορβηγία. Ή θα μπορούσαμε να επιμείνουν ναι, οι κάτοχοι να έχουν μακρόχρονη δράση ε, στο τομέα, έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάποιοι ε, να δυσδύουν. Και Έχουμε μια μεγάλη γκάμα. Κάθε πρόβλημα που άκουσα να αναφέρεται εδώ σε σχέση με τις ε, βιβάσιμες ελευτικές παραχωρήσει μπορεί να αντιμετωπιστεί ανάλογα με το πώς θα καταρτιστούν. Ε, βέβαια, υποπτευούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν και τόση διάθεση να το πράξουν γιατί θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη. Και αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια ε, αυτά θα κατηγορηθούν, όχι οι Βρυξέλλες. με πολλούς τρόπους ε, είναι μία από τι μεγαλύτερε πράξει περιφερειοποίησης που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Κάθε κράτο βαλός πρέπει να συστήσει ένα σύστημα που θα ταιριάζει με τι δυστικέ του εθνικέ προτεραιότητε. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι αυτό το δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, εκτός ε, και αν το θέμα της τη ελευθερικής ικανότητας μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώ. Όμω, νομίζω ότι η εισηγήτρια έχει παρουσιάσει κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις ε, να έχουμε σαφή ορισμό τη και δεχόμαστε ε, με ποιο τρόπο, με ποια μέτρα θα το μειώσουμε αυτή. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να το δούμε για την περιφερειοποίηση. Όλοι είναι υπέρ, αλλά όπως το κατανοώ εγώ, όπως ε, ερμηνεύω τον κανονισμό της Κομισιόν, η περιφερειοποίηση υποτίθεται ότι θα είναι μια διαδικασία από κάτω προ τα πάνω. Δεν θα προσπαθήσει η Κομισιόν να πει ποιο θα κάνει τι, αλλά η Κομισιόν λέει θέλουμε την αποκέντρωση, θέλουμε να σταματήσει η μικροδιαχείριση, αλλά πρέπει να αναδυθούν κάποιοι φορεί ε, και θέλουμε αυτού του φορείς να αναδεικτούν που θα έρθουν εδώ και θα μα πούν θέλουμε να κάνουμε αυτό και θα ζητήσουν την έγκριση τη Κομισιόν. Και θα ε, λάβουν θετική αποδοχή. Αλλά τι θα γίνει αν δεν εμφανιστούν αυτοί οι φορείς ε, και ε, χάρη ε, στη Σκοτία ε, ε, αναφέρθηκε στο να δοθεί κάποια εξουσία σε κάποιου ε, πιο μικρού φορεί, όπω μπορεί, παραδείγματο χάρη, σε άλλα κράτη-μέλη μπορεί να μην υπάρχουν φορεί που να νιώθουν έτοιμοι να αναλάβουν το βαθμό τη ευθύνη που αναφέρεται εδώ. Και όταν ε, αναλάβουν τι ευθύνε, τότε αυτοί που λαμβάνουν τι αποφάσει, ξέρετε, θα κατηγορηθούν. Ε, όχι οι Βρυξέλλε, Λοιπόν, ε, εγώ ανυπομονώ το ε, Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, Πατριωτικό Κόμμα να κατηγορηθεί. Ε, περιμένω αυτή τη μέρα, όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν κανόνες και θα παρέχουν και ένα δίκτυο ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάποιες βασικές αρχές που θα ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η περιφερειοποίηση θα αναπτύσσεται με πιο βραδείς ρυθμούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, mm, Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα και εγώ να επενέσω την πολύ καλή δουλειά της Ουλρίκε Ρόντουστ. Την ευχαριστούμε και την συγχαίρομαι για την εξαιρετική δουλειά. Τώρα, επί της ουσίας, εφιστώ την προσοχή σας στα δεδομένα μας. Η Ουλρίκε αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων. Και όποιος επιχείρησε να μελετήσει σε βάθος το πρόβλημα των στατιστικών δεδομένων συνήθως κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, δεδομένα ή σε επίπεδο οργανισμών που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ε, πολιτική αλίας. Οπότε το θέμα των δεδομένων γίνεται κύριο θέμα, αλλιώς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποθέματα. Πολλές φορές προσπάθησα να κάνω ερώτηση στην Κομισιόν για δεδομένα για διάφορα είδη και δεν υπήρχαν δεδομένα. Οπότε είναι φυσική πορεία αυτή που πρέπει να ακολουθήσουμε ε, σε σχέση με τα δεδομένα. Πρέπει να τα ζητήσουμε ή θα πρέπει να ζητήσουμε από τους αλληλείς να μας τα δώσουν. Αλλά δεν θα μας τα δώσουν αν το σύστημα υποβολής αναφοράς δεν είναι ενιαίο, ενοποιημένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ε, είναι παρόμοιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί μπορεί σε ένα κράτος μέλος να ε, χωρίζεται η ποσόστοση με τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε μια μέρα να πηγαίνει να ψαρέψει στα πλαίσια της ποσόστοσης ο αλιέας, ενώ την επόμενη μέρα πηγαίνει ως σκάφος αναψυχής. Ε, και την τρίτη μέρα χρησιμοποιεί τη βασική του ποσόστοση. Έτσι όμως εμείς δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ πώς χωρίζονται αυτές οι ποσοστώσεις και πώς γίνεται η υποβολή των εκθέσεων και των αναφορών αυτών. Και στο τέλος θα έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία κάθε κράτος μέλος θα παρουσιάζει τον αριθμό των ψαριών που ψάρεψε στα πλαίσια της ποσόστοσης, γιατί αν ξεπεράσουν την ποσόστοση θα φοβούνται ότι θα έχουν επιπτώσεις και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο όπου χωρίζονται κεντρικά οι ποσοστώσεις αλλά αυτός ο επιμερισμός είναι αναξιόπιστος και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε σωστά στατιστικά στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι η μόνη λύση είναι να ε, έχουμε τον ίδιο τρόπο επιμερισμού των ποσοστώσεων Μιλώ για κάποιες βασικές αρχές, δηλαδή δεν ε, αναφέρομαι σε, στα είδη. Πρέπει να χωρίζουμε τις ποσοστώσεις με βάση συγκεκριμένες γενικές αρχές. Τώρα για την απαγόρευση των απορρίψεων, ε, αυτό είναι ένα θέμα που βρίσκει σύμφωνους όλους και θα πρέπει να θεσπιστεί το ταχύτερο δυνατόν γιατί είναι σκανδαλώδες να υπάρχουν τα παρεμπίπτοντα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμάστε όμως ότι η απαγόρευση των ε, απορρίψεων που αναδεικνύεται ιδιαίτερα στα βιομηχανικά αλλιεύματα μπορεί να είναι μοιραία για ορισμένες ζων, περιοχές αλληλείας στη Βαλτική ή τη Μεσόγειο για παράδειγμα ή για ορισμένα είδη συγκεκριμένο που η βιομηχανική αλληλεία κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Αν λοιπόν θεσπίσουμε την απαγόρευση των απορρίψεων, θα δώσουμε το πράσινο φως στην, για την αύξηση της βιομηχανικής αλληλείας και στο τέλος θα καταλήξουμε σε χάος και σε παράλογες δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της Μεσογείου, γιατί εκεί θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά το θέμα. Να θυμάστε όμως ότι ορισμένα είδη στη Βαλτική επιβιώνουν όταν αλλιευθούν, αλλά απορρίπτονται με τρόπο φυσικό γιατί ε, κάποια είδη μπορούν να επιβιώσουν μέχρι το τέλος της περίοδου και μπορούν να γίνουν ένα εμπορικό είδος υψηλής ποιότητας. Όταν μπορούν να απορρίπτουν κάποια τέτοια είδη, δεν θα το κάνουν γιατί θα ε, προσπαθούν να ε, βελτιώσουν και να προστατεύσουν το περιβάλλον, από την άλλη ε, ακολουθούν κάποιες συνήθειες. Τώρα, για την, το, τα, νερά ηχθίδια, αν έχουν υψηλότερη τιμή, μειώνονται οι απορρίψεις. δεν θα θέλουν ε, θα, θα αυξηθούν οι απορρίψεις γιατί δεν θα θέλουν να μπει στον κατάλογο και να πληρώνουν για αυτά. Τώρα για τα βενθικά είδη, ή, τα πελάγια είδη και την πελάγια αλία, εκεί δεν έχουμε πολύ καλό έλεγχο των αλλιευμάτων, γιατί είναι λίγο τυχαία τα αλλιεύματα. Εδώ είναι σημαντικός ο αλιευτικός εξοπλισμός τι εργαλεία χρησιμοποιούν. Τέλος, το προτινόμενο ταμείο που θα διαχειρίζεται τις απορρίψεις, αυτό είναι πολύ καλή λύση πιστεύω, διότι για, θα, για κάποιες δραστηριότητες ε, θα αυξηθεί η, αξία των απορριπτωμένων ψαριών που δεν θα καταναλώνονται από τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να χρησιμεύουν για ηχθιάλευρα ή για τροφή για τα ψάρια. Τέλος για την α, περιφερειοποίηση, αυτό είναι θέμα πολύ σημαντικό επίσης και εδώ θα πρέπει οι απορρίψεις ε, να λύνονται από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια στις διάφορες περιοχές, γιατί αυτά τα συμβούλια έχουν την καλύτερη γνώση επιτοπίως και μπορούν να βοηθούν στην νομοθετική διαδικασία και στη θέσπιση κανονισμών και είναι υπόλογα ε, των για τις πράξεις τους. Και βέβαια όταν κάποιος είναι υπεύθυνο και υπόλογος, τότε τα νομοθετήματα και οι κανονισμοί δεν θα είναι εικονικά, αλλά θα εδράζονται σε μια σωστή πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Γέρου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ρόντουστ για την εκθεσή της. Πιστεύω ότι πραγματικά έχει κάνει αξιοσημείωτη προσπάθεια να συμπεριλάβει όλες τις πτυχές Εγώ από την στιγμή που άρχισα να συμμετέχω σε αυτό το κοινοβούλιο έχω μπορέσει να ακούσω και την Επιτροπή αλλά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν ορισμένε πτυχέ που θα προτείνει η Ισπανική Αντιπροσωπεία γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο. Ω είναι λογικό. Και βέβαια ούτε βρισκόμαστε και στην ε, στιγμή ε, κατά την οποία θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις. Όμως θέλω να πω ότι ε, αυτό το έγγραφο προκύπτει κατόπιν μεγάλης προσπάθειας και κατόπιν μεγάλης συνεργασίας. Μας ζήτησε η συγκεκριμένη συμμετοχή μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμείς ε, από την πλευρά της Ισπανικής Αντιπροσωπείας συνεισφέραμε με τις προτάσεις μας. Πέρα λοιπόν από τον ενθουσιασμό που μπορεί να μας ε, προκαλεί ένα έγγραφο, ε, το οποίο είναι υπό την ευθύνη των ε, βουλευτών ε, στην περίπτωση αυτή των Ισπανών πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για μια καινούργια κατάσταση. Από τη στιγμή της θέσεως ισχύς συνθήκης Λισαβόνας το Κοινοβούλιο μπορεί για πρώτη φορά να συμμετέχει στον προσδιορισμό της κοινής πολιτικής. Και αν είναι δύσκολο και μέχρι τώρα δεν έχει συζητηθεί ένα τέτοιο θέμα τα τελευταία 30 χρόνια ακόμη πιο δύσκολο θα είναι κάποιος ε, βουλευτής ε, ε, να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο φοιτηρίας αυτό. Και θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε κάποια σύγκριση που έκανα και με προτάσεις άλλων συναδέλφων. Και πράγματι, υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχουν σημαντικές διαφοροποίησεις. Γιατί εμείς που υπερασπίζουμε τα κοινωνικά ε, συμφέροντα, τα περιβαλλοντικά συμφέροντα, και μας, ε, μας ενδιαφέρει να περισπίσουμε τα συμφέροντα αυτά, αλλά μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε και ζωντανή αυτή την ε, αλία και να έχουμε και ένα βιώσιμο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλους ε, τους παράγοντες και τους κοινωνικούς και τους οικονομικούς και τους περιβαλλοντικούς. Και έτσι λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι η Ισπανία ε, μπορεί να έχει μια καθολική ε, προσέγγιση ε, και μπορεί να προσφέρει και προϊόντα πρώτης ποιότητας. Εμάς μας ενδιαφέρει να το δούμε το θέμα με πιο αντικειμενικό τρόπο και γι' αυτό πρέπει να δούμε τα θέματα που προκαλούν μεγαλύτερη αμφισημία, που είναι τα πιο επίμαχα. Πρέπει να τα δούμε βάσει περισσότερων πληροφοριών και θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός χαρακτήρας, ε, να έχουμε επιστημονικές μελέτες και μελέτες αντικτύπου για κάθε ελίευμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στη συνέχεια όταν θετείται κάποιο σχέδιο θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Τώρα να προχωρήσουμε στην... Ε, μεταρρύθμιση έχοντας κατά νου ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον κλάδο και κυρίως τους ε, αλληλείς ε, μικρής κλίμακας. Ε, την αλία μικρής κλίμακας, γιατί αυτοί με τη στάση τους μπορούν να συνεισφέρουν στο να έχουμε όσο το δυνατόν βιώσιμη αλία. Το πλαίσιο για την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ευέλικτο, πρέπει να ειδωθεί από διαφορετικό ε, από διαφορετική σκοπιά. Η λύση που προτείνεται εδώ είναι για τη βιομηχανική αλία και όχι τόσο για την αλία μικρή κλίμακα. Έτσι λοιπόν πρέπει να ε, το δούμε αυτό το θέμα και με τις ε, επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου και επίσης πρέπει να υπάρχει και στο δυνατό μέγιστη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους ρεαλιστικούς στόχους, αυτούς τους εφικτούς στόχους. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό για την υδατοκαλλιέργεια και στη βιομηχανική αλλά και σε παραδοσιακή κλίμακα. Εμάς ε, θα μας ενδιαφέρει να αναφέρεται αυτό το στοιχείο με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, όταν κάνουμε λόγο για το αν ε, έχει γίνει πρόοδος ή όχι έχει γίνει πρόοδος, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως φυσικά δεν αρκεί η πρόοδος αυτή. Και το να είμαστε κατά είναι να προχωρήσουμε στην πολιτική των των αλλιευμάτων είναι κάτι θεμελιώδες. Και επίσης, ε, γι' αυτό το λόγο είναι θεμελιώδες από τη δική μας σκοπιά να δούμε τα προβλήματα ε, ανά αλλιεύμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Και τώρα αναφέρουμε στις μεταβάσιμες, στις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από αυτά τα ελεύματα για τα οποία ήδη υπάρχει μια ποσόστοση και με ευελιξία να μελετήσουμε τη δυνατότητα να εισαγάγουμε αυτές τις ποσοστώσεις και να τις μεταφέρουμε μεταξύ των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα πρόληψης, κύρωσης, τα μέτρα διοικητικού ε, χαρακτήρα, νομικού χαρακτήρα νομίζουμε ότι είναι σημαντικά. Πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε και στην δημιουργία των ε, επιστημονικών και τεχνικών μέτρων έτσι ώστε να έχουμε μία πιο υπεύθυνη και βιώσιμη αλία αλλά και καλλιέργεια. Και τέλος, να πω ότι είναι προφανές ότι όλη αυτή η μεταρρυθμίση δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε επαρκείς ε, οικονομικούς πόρους. Και αυτοί οι οικονομικοί πόροι θα έπρεπε να μεταφραστούν και σε μια οικονομική μνήμη. Δηλαδή δεν μπορούμε ε, με αντικειμενικό και ρεαλιστικό τρόπο να προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουμε μια κατάλληλη διάγνωση, αν ε, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τους στόχους και αν δεν έχουμε και τους απαιτούμενους ε, οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση. Έτσι λοιπόν κλείνω λέγοντας πως ε, οι, εμείς ε, οι ε, είμαστε υπέρ μιας μεταρρύθμισης της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής που να διατηρεί αυτούς τους στόχους, το κοινωνικό, το οικονομικό και το περιβαλλοντικό σε θέση προτεραιότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την κυρία Ρόντου, στην εισηγήτρια, η οποία ανέδειξε όλα τα βασικά σημεία και έκανε και προτάσεις. Επί αυτών συζητούμε τώρα. Ή ο κλάδος της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιορισμένο βαθμό είναι παγκόσμια ανταγωνιστικός και ε, λειτουργεί σε περιορισμένες ε, συνθήκες ε, γι' αυτό σε περιορισμένο βαθμό ε, και ε, χωριστά αναλαμβάνονται δράσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για να προστατεύσουμε και τους, την ελία μικρής κλίμακας και την μελάγια αλία και την παράκτια αλία και να τις διατηρήσουμε όλες εν ζωή στην Ευρώπη. Κυριολεκτό εδώ. Τα αποθέματα λοιπόν θα πρέπει να ε, έχουν την σωστή βιομάζα σε σχέση με τη θνησιμότητα και θα πρέπει να ορίσουμε και χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία θα λαμβάνουμε μέτρα ούτω ώστε να έχουμε βιώσιμη απόδοση ε, μακροπρόθεσμα. Για τις απορρίψεις δεν μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε στο παρελθόν. Όλοι συμφωνούμε, γιατί εδώ έχουμε κατασπατάληση βιομάζας που αλλιεύτηκε, ε, πήγε στο, έφτασε στο σκάφος, επέστρεψε στη θάλασσα και ε, χρησιμεύει για τροφή των γλάρων ή οτιδήποτε άλλο. Ε, αυτά πολλές φορές είναι ωραία εδόδημα ψάρια. Και ξέρουμε ότι οι ποσοστώσεις ε, ε, επιμερίζονται με βάση τις παραχωρήσεις και πολλές φορές γίνονται πολύ περίεργα πράγματα. Θα πρέπει βέβαια οι αλληλείς να πιστούν ε, να συνεργαστούν για την απόρριψη και την απαγόρευσή τους. Πρέπει να πιστούν ότι αν τηρήσουν την απαγόρευση θα τους ωφελήσει αυτό. Γιατί αν ε, επιμερίζονται όλα στις ε, ποσοστώσεις, ε, ό,τι εκφορτώνεται και ό,τι πάει απάνω στο πλοίο, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η πρακτική τα προηγούμενα χρόνια και πόσα καλά εδόδημα ψάρια γύρισαν στη θάλασσα. Πρέπει να έχουμε στοιχεία, να το βρούμε αυτό το πράγμα. Πόσο, 10 τόνοι, 10 χιλιάδες τόνοι ε, μπακαλιάρο για παράδειγμα που για κάποιους λόγους ε, ε, πήγαν στην απόρριψη. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Επίσης η θνησιμότητα των ψαριών και τα αίτια της. Επίσης τα νεαρά ηχθίδια και η ποσόστοση. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σε ποιο βαθμό και πώς θα υπολογίζεται. Και ποιος θα το ελέγχει αυτό το πράγμα εντάξει, μιλάμε για απλοποίηση, για μείωση της γραφειοκρατίας κλπ. Και τα έχω πει και εγώ ίδιο στο Κοινοβούλιο, έχω βγάλει λόγο για αυτά τα θέματα. Πρέπει όμως να σκεφτούμε πολύ συγκεκριμένα πώς θα λειτουργήσει το καινούργιο σύστημα και πώς θα θέσουμε όλα αυτά τα θέματα υπό έλεγχο. Τώρα για την κατανομή, των επιμερισμών των ποσοστώσεων στα κράτη-μέλη, ε, το βασικό θα είναι η συμφωνία του 82 με τη σχετική σταθερότητα και μπορούμε τα επιμέρους να τα ρυθμίσουμε και να τα συζητήσουμε. Τώρα, για τις ε, μεταβιβάσεις μιας αλλιευτικές ε, παραχωρήσεις, ε, θα πρέπει εδώ να λαμβάνουμε υπόψη μας όχι το πρόσωπο αλλά το αλλιευτικό σκάφος και από κοινού θα πρέπει να συσκεφτούμε και να δούμε πώς θα συνεχίσει στο μέλλον να λειτουργεί μια επιχείρηση κάποιος ας πούμε που κάνει παράκτη αλληλεία και συνταξιοδοτείται. Τι θα κάνει ο νέος αλλιέας. Μπορεί να ε, πάρει όλο το αλλιευτικό σκάφος και τα εργαλεία, αλλιεύση, τα αλλιευτικά εργαλεία κλπ. Και να τα λειτουργεί. Ε, αυτό θα πρέπει να το δούμε και από το Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Να υπάρχει μια χρηματοδότηση ούτως ώστε ένας νέος αλιέας να μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Ε, τώρα, για το χειρισμό των ε, ποσοστώσεων, συμφωνώ εδώ με την εισηγήτρια. Για τις αλλιευτικές ε, ικανότητες, την αλλιευτική ικανότητα, βεβαίως παίζει ρόλο κινητήρας, αλλά και τα αλλιευτικά εργαλεία στο μέλλον και αυτά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, πολύ καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να διαθέσουμε όμως επενδύσεις, γιατί δεν μπορούμε να διευρύνουμε αενάως τις ε, ε, επιχειρήσεις ε, ή να τους πούμε ότι με συγκεκριμένα εργαλεία θα πρέπει να αλλιεύεται συγκεκριμένα είδη. Ενώ θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα τα σκάφη. Τώρα, για τα ΡΑΚ, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, για το, το, τις ρυθμίσεις, θα πρέπει να, και οι καταναλωτές και οι εργοδότες εργαζόμενοι ε, να συμμετέχουν, η οικονομία και η εμπειρία των επιστημόνων επίσης είναι σημαντική. Η καλλιέργεια, θα παίξει μεγάλο ρόλο και όταν μιλάμε για παρεμπίπτοντα αλλιεύματα που εκφορτώνονται όλα. Ε, αυτά είναι ε, πηγή λευκομάτων που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί πρακτικές λύσεις που μπορούμε να βρούμε. Ε, μίλησα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τώρα για τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο χωριστά να τα ξαναδούμε, χρειάζεται αυτό. Δεν μπορούμε όλα να τα ε, βάζουμε στον ίδιο κουβά. Καμιά φορά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και όταν έχουμε ας πούμε εφαρμοστικές διατάξεις 116 σελίδων με πολλές λεπτομέρειες και ορισμούς, ε, δεν θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ε, ιδιαιτερότητες σε περιφερειακό επίπεδο. Καλό είναι λοιπόν να τα ξαναδούμε όλα αυτά και συμφωνώ ε, με την εισηγήτρια σε σχέση με αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ κύριο Σαρσένης. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγητρία για την πολύ καλή δουλειά που έκανε για αυτό το έγγραφο. Θα συμφωνούσα σε πολλά σημεία. Έχετε λοιπόν τη γενική μου υποστήριξη, αλλά θα είδα Ήθελα να δω πιο ισχυρή διατύπωση σε δύο σημεία. Συγκεκριμένα στην πρόταση 16, στην ε, ιδέα των ευέλικτων ποσοστώσεων, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρονται οι μη χρησιμοποιημένε ε, ποσοστώσει ε, από χρόνο σε χρόνο. Νομίζω ότι αυτό έχει μια λογική στα μαθηματικά αλλά στην ε, βιοπικιλότητα δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα και το ίδιο ισχύει και για τα υποθέματα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει πάντα να λεβούμε βάσει των επιστημονικών δεδομένων και φαίνεται λογικό να μπορούμε να μεταφέρουμε ό,τι δεν αλλιεύσαμε το 2012 στο 2013. Αλλά μπορεί η πρόσθετη πίεση που να έχει προκύψει ε, βάσει ορισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών ε, να έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες. Έτσι λοιπόν αυτή η λογική δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Πρέπει ε, πάντοτε να βασιζόμαστε στα επιστημονικά στοιχεία και τα επιστημονικά στοιχεία λαμβάνουν υπόψη την ε, ποικιλομορφία ε, την μεταβλητότητα των φυσικών συνθήκων που μπορεί να έχουν συνέπειες και στα αποθέματα. Και επίσης, όπως ε, και με τον κύριο Μιλάνα και με πολλούς άλλους συναδέλφους, ε, θα ήθελα να πω και εγώ με σαφήνεια πόσο σημαντικό θα ήταν η μεταρρύθμιση αυτή να είναι αποτελεσματική και να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και να μας επιτρέψει να έχουμε και αλείς αλλά και ψάρια στις θάλασσές μας τα επόμενα δέκα χρόνια και να έχουμε αποθέματα. Συμφωνώ ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη Μεσόγειο. Θα ωφελήσει όλα τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιστεύω ότι τον έχουμε αυτές τις επαγγελματικέ περιοχές που θα επιλέγονται από κάθε κράτο μέλο και θα επιλέγονται με διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και τους ελλεί και επιλέγουμε να μην ελεύουμε εκεί και γύρω από εκεί μπορούμε να ελεύουμε όπως ε, έχει δείξει η εμπειρία ε, περιγαλύτερες με λιγότερη προσπάθεια νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα κρίνουν σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης το αν ε, θα μείνουν αλείς. Γιατί θα κρυθεί και από το αν θα μείνουν ψάρια εκεί. Αυτά και πάλι σας ευχαριστώ για την ε, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Μιράντα. Ευχαριστώ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η κοινή ελευτική πολιτική ακολουθούσε τα κριτήρια της διακυβέρνησης, δηλαδή τη λήψη αποφάσεων ε, βάσει των καλύτερων ε, γνωμοδοτήσεων των επιστημονικών, όπως συμμετέχουν ενεργά για τα διαφορεμένα μέρη και έχουμε και μια μικροπρόθεσμη προοπτική η επιτυχία της διαχείρισης, δηλαδή η αποτυχία της σημερινής διαχείρισης οφείλεται στο ότι υπήρχε έλλειψη ευθύνης, ανάληψη ευθύνης ε, σε τοπικό, σε περιφερειακό σε εθνικό, κρατικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε έλλειψη ε, ανάληψης ευθύνης, υπήρξε έλλειψη καλής διαχείρισης ε, των μέτρων προστασίας ε, και των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών μέτρων. Γι' αυτό η έκθεση της κυρίας ε, Ρόντουστ ε, που θέλει να αμφισβητήσει ε, τη μεταρρύθμιση και θέλει να παρουσιάσει μία μεταρρύθμιση πιο φιλόδοξη αφορά και συγκεκριμένες θέσεις για ορισμένα ελεύματα. Αν δούμε ένα κριτήριο που θέτει η κυρία Ρόντου στο σημείο 22 για τον ορισμό του μικρού αλιέα, είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτό το πλαίσιο η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν Μάλλον είναι απογοητευτικό το ότι δεν γίνεται αναφορά στην διαφορετική μεταχείριση της ε, μικρής αλίας ε, ούτε ε, στους βιοτέχνες αλής και έχουμε κάποιες περιοχές όπως τη Γαλλικία, τη δική μου, που έχουμε 200.000 άτομα που εξαρτώνται από αυτή την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και είναι βιώσιμο ουσιαστικά δεν χρειάζεται τίποτα μεγαλώνουν μόνοι τους αυτοί οι οργανισμοί και παρέχουν ε, και δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Εμείς υποστηρίζουμε μία θέση διατήρησης ε, των πόρων ε, και θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα αποθέματα του πληθυσμού, πρέπει να τα προστατεύσουμε, πρέπει να είναι καθαρά τα ύδατα για να επιβιώνουν τα ψάρια, αλλά επερασπίζουμε και μία πολιτική διατήρηση των ε, αποθεμάτων. Γιατί ε, δεν μπορούμε να έχουμε ελευτική πολιτική αν δεν υπάρχει και πολιτική διατήρηση των πόρων αυτών των ελευτικών περιοχών. Πριν μία εβδομάδα ε, μου είπε ένας ε, ψαράς ο παππούς μου και ο πατέρας μου ε, ήταν αλής, εγώ είμαι αλίας και ο γιος μου ετοιμάζεται να γίνει και έχουν ένα σκάφος και χρησιμοποιούν οικολογικά εργαλεία. Ε, την πραγματικότητα που βλέπουμε στην Γαλλικία, στην Καντάμπρια, στις ε, της Γαλλίας, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και σε άλλους ε, τόπους ε, πρέπει να δοθεί μια απάντηση στην Επίτροπο και στον Κομισιόν και γι' αυτό ε, η κυρία Ρόντους, συγγνώμη αλλά δεν μας ακούτε τώρα, θέλουμε ε, να σημαίνει το εδώ. Υπερασπίζεστε ένα διαφοροποιημένο σύστημα και το χάρη μπορούμε να δούμε τη χρήση των ελευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Και υπάρχει μεγάλη εμπειρία για αυτό το θέμα σε ορισμένα κρατημέλη. Σε αυτό το πλαίσιο για τις μεταβιβάσιμε ποσοστώσει θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε την ε, δυνατότητα, τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα προστασίας που θα μπορούν να προστατεύσουν τις, ε, την παραδοσιακή αλία να αποκλείεται από τα τάκια τις ποσοστώσεις. Και αυτό προτείνει ο κλάδος. Γιατί ε, τελικά Οποιαδήποτε πολιτική προτείνουμε εμεί ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν, από τα κράτη-μέλη, ε, αν δεν ε, συμμετέχει και ο κλάδο, δεν θα διαμορφώσουμε μια σωστή πολιτική. Και θέλω να αναφερθώ και στα προγράμματα διτοκαλλιέργεια. Εγώ προέρχομαι μια χώρα όπου έχουμε εκτατική υδατοκαλλιέργεια. Είναι πράσινη, είναι οικολογική, είναι βιώσιμη και δεν. Ε, ε, είναι υπέρ ο τομέα να δημιουργήσει μια εντατική υδατοκαλλιέργεια με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μελλοντικό ταμείο, ναι, θα έπρεπε να χρηματοδοτεί την υδατοκαλλιέργεια, αλλά εκτατική, όχι εντατική, που να επικεντρώνονται οι πόροι στα χέρια ορισμένων και να μην είναι ε, και ε, βιώσιμη γιατί έχουμε διάφορα είδη ε, παραδείγματο χάρη δεδοκαλλιέργεια που είναι βιώσιμα έχουμε το χάρη περιπτώσει βιώσιμη δεδοκαλλιέργεια στις ακτέ τη Γαλλικία. και εμεί κάτι τέτοιο θέλουμε να περασπίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ρόσπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι είπαν ήδη πάρα πολλά πράγματα που δεν θέλω να τα επαναλάβω. Πρώτα θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ρόντους για την εξαιρετική δουλειά, δουλειά σε βάθος, σε εύρος, κάνατε πολλή δουλειά, ευχαριστούμε. Και βεβαίως με πολλές από τις καλές σας προτάσεις συμφωνώ. Τώρα, εγώ θα μιλήσω μόνο για την υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει να προωθήσουμε την οικολογική και την βιώσιμη ε, υδατοκαλλιέργεια, η οποία θα αποφέρει τα περισσότερα. Εδώ δεν μιλάω μόνο για την Πορτογαλία, την Ισπανία ή τη Δανία, ε, τη δική μου χώρα, που είναι παράκτιες χώρες. Μιλάω για χώρες περίκλειστες, όπως την Αυστρία, με μικρές λίμνες, μεγάλες λίμνες ή την Ουγγαρία κλπ. Θα πρέπει και εκεί να ρυθμίσουμε το ζήτημα πάνω στη βάση των και να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές, ε, όπως λέτε πολύ σωστά, να τηρούν τους κανόνες ευζοίας των ζώων, ε, τους περιβαλλοντικούς κανόνες, να είναι πάνω σε σωστά γερά θεμέλια η υδατοκαλλιέργεια η οποία είναι ανανεώσιμη μορφή και μπορεί να γίνει ε, βιολογική ή οικολογική και να ε, λειτουργήσει έστω στη βάση. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δρομεύα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί της ουσίας ακούσαμε ήδη πάρα πολλές παρεμβάσεις ε, που φαίνονται λογικές κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα όμως και εγώ να προσθέσω κάποια πράγματα σε σχέση με κινδύνους ε, που ελοχεύουν κατά τη γνώμη μου στην ε, πρόταση μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ε, θα Ήθελα να συνοψίσω αυτούς τους λόγους. Ε, θα ξεκινήσω από τον στόχο της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να επανειεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας, ε, να έχουμε καλύτερη διατήρηση των αποθεμάτων, να μειώσουμε τις απορρίψεις, ε, να εγγυηθούμε βιώσιμη διατήρηση αποθεμάτων. Μάλιστα, η τίτλοι είναι εύκολη και η θεωρία το ίδιο. Το πρόβλημα είναι η πράξη. Εγώ θεωρώ ότι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόταση που θα μπορούσε να προκύψει από το σχέδιο της ε, κυρίας Ρόντους το συνεπάγονται εξίσου ε, μεγάλους ε, κινδύνους. Τονίζουμε τι είναι εύκολο να υποπτεύσουμε και δεν αφιερώνουμε καθόλου, αφοσιωνόμαστε καθόλου στα πρακτικά προβλήματα, δηλαδή στα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε και πώς να τα χρησιμοποιήσουμε για καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων. Φυσικά είναι περίπλοκο το ζήτημα. Φυσικά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην απαγόρευση της απόρριψης, μεταβιβάσιμε ποσοστώσεις, μεταβιβάσιμε παραχωρήσεις. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι και θα πρέπει να αποτελέσει αυτή η λύση τμήμα μιας ε, σφαιρικότερης ε, πολιτικής ε, και ακριβώς σε αυτό έγκυται το πρόβλημά μου. Έχοντας ακούσει τη συζήτηση θεωρώ ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις αλλά δεν έχουμε σφαιρική πρόταση Ε, το εύκολο είναι να επιτίθενται κάποιοι σε εισαγωγικά, δηλαδή να υποπτεύουν τις ηχθειοκαλλιέργειες, γιατί είναι μικρές εκμεταλλεύσεις, εύκολα μπορεί να πάει ο επιθεωρητής επιτόπου να ελέγξει ακριβώς τι γίνεται, πολύ ευκολότερα σε σχέση με την απόρριψη από το σκάφος στα ανοιχτά οποιοδήποτε είδους ψαριού δεν χρειάζεται αλλαγή των τεχνικών ικανοτήτων των σκαφών, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την μείωση των απορρίψεων. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η ιδανικότερη λύση και για τις ηχθειοκαλλιέργειες πιστεύω ότι ο στόχος μας δεν θα έπρεπε να ε, θέλουμε να αυξήσουμε την εκτροφή εγκλωβισμένων ηχθείων. Θα πρέπει στο φυσικό τους βιότοπο να εκτρέφονται τα ψωρία. Γι' δεν, αυτός δεν είναι δευτερεύον στόχος. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πρωτεύον. Σε σχέση λοιπόν με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο της κυρίας Ρόντουστ, πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκυται στην λανθασμένη μετατόπιση των κονδύλιων, λανθασμένη επανειεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Αυτό με φέρνει και σε ένα τελευταίο σημείο σε 15-20 χρόνια πώς θέλουμε να διαμορφωθεί η αλληλεία, ποιος ε, θέλουμε να ψαρεύει σε 20 χρόνια ή για να το πω ακόμη απλούστερα ποιος δεν θέλουμε να ψαρεύει σε 20 χρόνια. Πρέπει να ληφθούν αυτές οι δύσκολες ε, πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες ε, και πλήττονται αυτοί που αξίζουν περισσότερο από όλου την υποστήριξή μας, ε, οι αλληλείς ε, δηλαδή. Ε, θα προσπαθήσω να μετατρέψω αυτή μου τη σκέψη σε συγκεκριμένε τροπολογίες, αλλά σας παρακαλώ να έχετε το νου σας, να κοιτάζετε το δάσος και όχι να εστιάζετε στα δέντρα Το δάσους. Ευχαριστούμε κύριε Ρομέντα. Η κυρία Πατρέων Εύεσε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, είναι πλεονέκτημα ε, να μιλάω από τους τελευταίους, ε, διότι μπορώ να περιοριστώ σε κάποιες ιδέες μόνο που μου φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν αναφερθεί. Θα επαναλάβω ελάχιστα πράγματα μόνο για να τα τονίσω. Αρχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Δεν θέλω να χάσω χρόνο, θέλω μόνο να τονίσω κάποιες σημαντικές κατεμεύτυχες του ζητήματος αρχίζοντας από τη σημαντική διάκριση ανάμεσα στην βιομηχανική και την ερασιτεχνική αλία. ούτω ή άλλως ανέκαθεν μας απασχολούσε αυτό το θέμα και μας απασχολεί ακόμη περισσότερο ε, στη νέα έκθεση, κυρίως η πρόταση 22, γιατί αναφέρονται εκεί συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό με απασχολεί, διότι... Στι πολλαπλέ συζητήσει που έχουν ήδη διεξαχθεί για αυτό το θέμα, είχαμε όλοι πει με σαφήνεια πω ε, ο ορισμός θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από ευελιξία για να είναι δίκαιη η λύση που θα βρεθεί τόσο για τον Βορρά όσο και για τον Νότο. Δεν ξέρω ως εκ τούτου σε ποιο βαθμό θα είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε έναν ενιαίο ορισμό που θα ισχύει από το Βορρά μέχρι και τον Νότο της Ευρώπης για αυτού του είδους ε, την αλία χωρίς ε, να προβλέψουμε αντικειμενικά κριτήρια, κριτήρια στάθμισης. Και το πρόβλημα τίθεται όχι μόνο σε σχέση με τον ορισμό, είναι προφανές, αλλά και σε σχέση με τις επιπτώσεις. Είχαμε καταλήξει στην εξή συνένεση, ε, ότι χρειαζόμαστε διαφοροποιημένο καθεστώς για την αλία μικρής κλίμακος. Ε, αυτό το διαφοβροποιημένο καθεστώς αγγίζει πολλούς κλάδους και θα αναφερθώ σε κάποιους μόνο. Ε, οι μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις, παραδείγματο παραδείγματος χάρη, πώς θα γίνει αυτό στην περίπτωση της ε, μικρής ε, κλίμακος αλίας. Πώς θα διατηρηθούν αυτές οι ποσοστώσεις. Εγώ θα ήθελα η διαχείριση των ποσοστώσεων να είναι ένα σύστημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την βιομηχανική ελεία. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ε, στην πράξη αυτό το σύστημα για την ε, αλεία μικρή κλίμακα. Τώρα για τι αλλιευτικέ ε, περιοχέ, πάλι για την ραστεχνική ελεία, μπορούμε να επιδιώξουμε τη διαφοροποίηση, αλλά σε τι θα ωφελήσει. Το ίδιο και για τις επιδοτήσεις. Το σχολιάσαμε προηγουμένως αντιλαμβάνομαι ότι η βιομηχανική αλληλεία δεν μπορεί να διοχετεύει οπουδήποτε τα ε, κονδύλια ε, της Ένωσης ε, και να ανταπορροφούν κάποιες επιχειρήσεις που στη συνέχεια αλλάζουν δραστηριότητα και κλείνουν, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για την μικρή κλίμακα αλληλεία. Στην τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο εγκρίναμε μία, ένα ψήφισμα σε σχέση με την πολυτροπικότητα της αλείας και εκεί ακριβώς εστιάζαμε την προσοχή μας στη μεγάλη στην ποικιλία, αν θέλετε, παραδοσιακών προϊόντων που προάγει η τεχνική ε, αλία. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω ε, στην εισηγήτρια μας να συμπεριλάβει αυτό το θέμα στην ε, έκθεσή της. Ε, το, αυτό της πολυτροπικότητας. Δηλαδή πέρα από αυτό υπάρχει και το θέμα της αίρεσιμότητας. Ε, θεωρώ παρόλα αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αιρεσιμότητα. Δηλαδή, είναι θετική διάκριση υπέρ αυτού που εφαρμόζει ε, αγαστέ πρακτικέ. γιατί έτσι, αν θέλετε, οι αλληλείς και οι αλληλευτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνουν εταίροι μας στις επιθεωρήσεις και στους ελέγχους που θέλουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αν επικρατήσει αυτή η διακριτική μεταχείριση πέραν αυτών που εφαρμόζουν τις σωστές πρακτικές. Πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα του ορισμού ε, των ε, βιογεωγραφικών πώς ευαίσθητων περιοχών. Στην χαρτογράφηση αυτών των περιοχών, καθώς και του βυθού των διαφόρων θαλασσίων περιοχών, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο ως προς τον εντοπισμό των ευαίσθητων ζωνών, δηλαδή ζώνες, περιοχές όπου αναπαράγονται τα ψάρια και όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί ηχθιδίων. Αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να ληφθούν δεόντως υπόψη ούτως ώστε να χαίρουν ενός ε, κατάλληλου καθεστώτος προστασίας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Άλλα δύο σημεία θα σχολιάζω και θα κλείσω. Δεν είδα, αλλά α, ε, ίσως δεν το πρόσεξα κιόλας. Τέλος πάντων δεν έχω δει καμία αναφορά στις διάφορες νέες προτάσεις, της ε, εξόχους απομακρυσμένες ε, περιοχές. Ε, ενώ όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτών των περιοχών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αναγνωρίζουμε την ε, ιδιαιτερότητά τους Νομίζω ότι τουλάχιστον μία ε, συγκεκριμένη αναφορά σε αυτές ε, τις περιοχές και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κλάδος της αλίας αυτής της περιοχής θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ε, σε αυτή την έκθεση. Τέλος, η χθιοκαλλιέργεια. Μάλλον είδα το καλλιέργεια. Εγώ Δεν καταλαβαίνω πώς θα ένα, ένα μόνο περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο να ασχοληθεί με ε, ολόκληρη την υδατοκαλλιέργεια και την ηχθειοκαλλιέργεια που παρουσιάζει τόσε διαφορές από περιοχή σε περιοχή με ένα μόνο ρακ ε, θα καλύψουμε την υδατοκαλλιέργεια είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι στα γλυκά νερά, είτε είναι σε περίκληση περιοχή, είτε είναι στα ανοιχτά, είτε είναι για ψάρια, είτε είναι για μαλάκια. υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές που μου φαίνεται ότι για να ε, διατηρήσουμε την επιστημονική ακρίβεια και αξιοπιστία κατά την εκτίμηση των ε, ωφελών που μας προσφέρει η ιδεατοκαλλιέργεια δεν μπορούμε να βασιστούμε σε συμβουλές ενός ενιαίου δηλαδή γνωμοδοτικού συμβουλίου για ολόκληρη την ιδεατοκαλλιέργεια. Κατά τα λοιπά συγχαίρω την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε κυρία Πατράου Νέβες. Ο κύριος Δρέκη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους συνεχάρισαν την εισηγήτρια για την ε, ποιότητα της έκθεσης που κατέθεσε. Όντως, το επιβεβαιώνουμε και εμείς, είναι μια εξαιρετικά καλή απόδοση, ας το πούμε έτσι, δοθήσεις και της περιπλοκότητας του ζητήματος ε, που ε, συζητούμε και του αριθμού των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που προτείνουμε στη δική μας πρόταση. Δεν άκουσα να ζητεί κάποιο διευκρινή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε σημείο. Οπότε, ίσω ε, θα ήταν καλύτερο να ε, διατρέξω εντάχει κάποια σημεία που είδαμε ότι συμπεριέλαβε η συγγήτρια στην έκθεσή της και να σχολιάσω και κάποιες από τις παρεμβάσεις ε, των μελών της Επιτροπής. Ένα σημαντικό στοιχείο που ε, συγκρατούμε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Πρόκειται λοιπόν ε, την ε, νέα πολιτική για τις απορρίψεις σχετικά με την αρχή της επιλεξιμότητας Ο στόχος είναι να αποφύγουμε τις ε, απορρίψεις και όπως τόνισαν και όσοι σχολίασαν ε, ε, το θέμα θα ξέρουν ότι η πρότασή μας στην καρδιά της περιέχει αυτή τη διάταξη ακριβώς για να αποφύγουμε τις απορρίψεις. Μία άλλη ανησυχία που είχαμε εμείς ήταν με ποιο τρόπο να αποφύγουμε τις αναπόφευκτες ορισμένες, ε, τα αναπόφευκτα ε, ορισμένες φορές παρεμπίπτοντα αλλιεύματα παρά την επιλεξιμότητα, παρά οποιαδήποτε πολιτική μπορεί κάποιος να εφαρμόσει για να αποφύγει τις ε, τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα ή απλώς τα παρελιεύματα. Ε, ε, φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε θαλάσσιας λεκάνης. Φυσικά το χρειαζόμαστε αυτό για να βρούμε την σωστή ισορροπία, να διατηρήσουμε για να, αν θέλετε, να εκλείψουν τα κίνητρα απόρριψης για τους ίδιους τους αλλιείς το νέο σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δηλαδή πρώτον να μην δημιουργηθούν άλλα κίνητρα υπεραλίευσης άλλων ειδών, διαφορετικών ειδών, γιατί θα δημιουργήσουμε νέα προβλήματα έτσι. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία παράλληλων αγορών σε κάποιες χώρες. Ε, τα ηχθίδια ε, πολλούνται σε ορισμένες χώρες σε ιδιαίτερα ακριβές υψηλές τιμές, οπότε θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και έχουμε σημειώσει τις παρατηρήσεις σας και θα τις συζητήσουμε εδώ υπηρεσιακά. σε σχέση τώρα με την το αν η, τα TFC, ε, οι, οι μεταβιβάσιμες δηλαδή οι παραχωρήσεις είναι η λύση για οποιαδήποτε υπερβάλλουσα, πλεονάζουσα αλλιευτική ικανότητα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε. Κανείς δεν είναι ιδιαίτερα επιστημονικός. Ξέρετε ότι βλέπετε στα χαρτιά πάνω αριθμούς και στοιχεία και όλα φαίνονται επιστημονικά, αλλά δεν δίνεται μία πλήρης εικόνα σε καμία περίπτωση για την πλεονάζουσα αυτή ικανότητα. Και το λέω αυτό διότι κατά τη γνώμη μας ε, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό εφαλτήριο για τη νέα μεταρρύθμιση, δηλαδή τρόπους τεχνικής ε, καταμέτρηση, αν θέλετε, τη πλεονάσεως αλληλευτική ικανότητας που να είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με αυτούς που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Ε, μία άλλη διευκρίνηση που θα ήθελα να κάνω σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια είναι η εξή. Και πάλι εδώ δεν προτείνουμε οτιδήποτε δεσμευτικό. Κάποιοι από τους ομιλητές, αν δεν κάνω λάθος, είπαν δεν επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να μπλέκεται στο θέμα της υδατοκαλλιέργειας. Ε, θέλουμε τα κράτη-μέλη να ασχολούνται με αυτό, μα και εμείς αυτό προτείνουμε. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα ε, συνεχίσουν να είναι ε, οι κλειδοκράτορες και θα εισαγάγουν ένα σύστημα οικονομικών ε, και άλλων κινήτρων για ε, πρασίνηση, ε, βιώσιμη, πράσινη μάλλον βιώσιμη καινοτόμα υδατοκαλλιέργεια και σκεμμένα αποφύγαμε τον προσδιορισμό των επιμέρους ε, ειδών υδατοκαλλιέργειας γιατί δεν θέλουμε να είμαστε περιοριστικοί και ούτε θέλουμε να υπερβούμε αυτά που θα μπορούσαμε ή που θα έπρεπε να κάνουμε ε, με έδρα της Βρυξέλλες. Επάντως, η βιωσιμότητα του κλάδου ε, έχει την κέρια σημασία και γι' αυτό αναφερόμαστε στην υδατοκαλλιέργεια στην πρότασή μας. Θα διαβιβάσω την ε, πρότασή σας σε περί ευελιξίας ως προς τις ε, ποσοστώσεις, την πρόταση δηλαδή της ε, εισηγήτριας. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτή τη λύση για να διαπιστώσουμε αν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός για να διαχειριζόμαστε τις ποσοστώσεις και σε σχέση με το σοβαρότατο πρόβλημα των απορρίψεων, όπως όλοι γνωρίζουμε. Κάτι τελευταίο για το στόλο μικρής, ε, για το στόλους μικρής κλίμακας. Άκουσα από πολλούς να λένε ότι χρειαζόμαστε ειδικό ε, ε, τμήμα μέσα στον κανονισμό για αυτού του είδους του στόλους μικρής κλίμακας. Θα πω κάτι εδώ και πάλι φυσικά θα διαβιβάσω την ιδέα της κυρίας Ρόντου στην υπηρεσία μου ε, σχετικά με το αν ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα κριτήρια, πέρα δηλαδή από το μήκος ε, του σκάφους. Ε, θα το δοκιμάσουμε. Αλλά τούτου λεχθέντου θα σας πω ότι το έχουν δοκιμάσει το παρελθόν συνάδελφοί μου αυτό το σύστημα και μου είπαν ότι συνεπάγεται πολύ, πάρα πολύ δουλειά ο ορισμός της ερασιτεχνικής αλίας, σε μικρή κλίμακα Είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο. να καταλήξουμε σε ένα ορισμό για τα TFCs, ε, για τις μεταβάσιμες ε, παραχωρήσεις. Ε, δεν θελήσαμε να επιστρέψουμε σε λεπτομέρειες και μείναμε στις γενικές αρχές, διότι θέλουμε ρυθμιστικές αρχές να είναι οι αρχές που είναι εγκύτερες του στόλου μικρής κλίμακας σε σχέση με τις ευρύξελες Και πάλι εδώ θα πρέπει ε, να μεριμνήσουμε ώστε ο νέος κανονισμός να μην εμπεριέχει οποιαδήποτε στοιχείο που να αντιβαίνει σε αυτούς τους στόχους. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ε, περίπλοκο να αποπειραθούμε σε ένα βασικό κανονισμό, να καταλήξουμε σε ομοιόμορφες για όλους ε, λύσεις και σε γενικούς ορισμούς. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να το δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστούμε και για να τελειώσουμε τη συζήτηση, η κυρία Ρόντους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τα καλά και ευγενικά τους λόγια. Βέβαια, το έργο δεν είναι μόνο δικό μου. Συμμετείχατε κι εσείς λίγος πολύ. Κάναμε και ως Επιτροπή πολλές ακρο... ακροάσεις για το θέμα και η ομάδα εργασίας μου οργάνωσε πολλές ακροάσεις για το θέμα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι έχω καλή ομάδα, για να μην πω εξαιρετική ομάδα που με στήριξε. Γιατί μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό θέλω να πω ένα θερμό ευχαριστώ και εδώ σε όλους. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι έκθεση αυτό που συζητάμε, είναι μόνο έγγραφο εργασίας. Και αυτό το έγγραφο εργασίας θα είναι η βάση για, για μια καλή έκθεση. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους ήρθατε και είπατε τις απόψεις σας τις προτάσεις σας που θα οδηγήσουν ε, σε τροπολογίες ή μπορεί και να γλιτώσουν κάποιες τροπολογίες. Ο στόχος της μεταρρύθμισης ποιος είναι. Στο τέλος να έχουμε το αίσθημα ότι τα αποθέματα τα σπρώχνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και από άποψη οικολογική και από άποψη οικολογική. Να βοηθήσουμε την αλληλεία, να βοηθήσουμε όμως να ανανύψει και η θάλασσα και τα αποθέματα. Έχουμε λύματα σε πολλούς τομείς, πάντα σε δημόσιες εκδηλώσεις. Λέω ότι η παλιά αλλιευτική μεταρρύθμιση ήταν μια καταστροφή και εμείς όλοι μαζί τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει αυτό να επαφίεται σε μεμονωμένα πρόσωπα, γιατί κατά το παρελθόν το είδαμε πολλές φορές ότι πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβαν στα σοβαρά την ευθύνη και την αρμοδιότητα που είχαν. Κάποια κράτη δεν έκαναν σωστά τους ελέγχους που έπρεπε και ως Κομισιόν και ως βουλευτές εμείς πρέπει να επεξεργαστούμε ένα κείμενο που σε τελευταία ανάλυση θα πιέζει αυτούς τους ανθρώπους κάποια στιγμή να αναλάβουν με σοβαρότητα το έργο τους και την αρμοδιότητά τους. Γιατί δεν είναι 12 παρα 5, η ώρα είναι 12, φτάσαμε στη 12η ώρα και πρέπει να δράσουμε. Από τις ε, παρεμβάσεις σας που τις κατέγραψα όλες μία-μία, κατάλαβα λοιπόν ότι συμφωνείτε επί της αρχής να υπάρξουν κάποιες παρεκκλήσεις. Θα μου τα υποβάλλετε γραπτός και θα τα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου, γιατί ως επιτοπλίστων συμφωνούμε επί της αλλαγής και επί της ανάγκης να γίνεται η δουλειά μας σωστά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί από κοινού και ευχαριστώ για την αρρωγή σας. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και αύριο την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 6 τη ημερησία διάταξη, τροποποίηση του κανονισμού 1300 του 2008 για τη θέσπιση πολιτού σχεδίου για το απόθεμα Ρέγκας που κατανέμεται δυτικά τη Σκοτίας και για την αλία του υποθέματος αυτού. Ο κύριο Στίβενσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η δεύτερη αντιλογή απόψεων ε, για τον κανονισμό αυτό. Είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση την τελευταία φορά στην Επιτροπή Αλίας για αυτό το ζήτημα να σας ε, πω ποιες είναι οι προτάσεις μου για τα εκτιμώντας. Ε, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές, αλλά έχω ευθυγραμμίσει κάποιες από ιδέες ε, για να είναι πιο επαναγνωστές. Αναφέρομαι σε τρία κύρια άρθρα. Καταρχήν στο άρθρο 1. Διατηρώ την διατύπωση για τη γεωγραφική τοποθεσία του αποθέματος 6α βόρεια ε, ορίζεται με σαφήνεια και αναφέρουμε εκεί που, ακριβώς όπου εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο. Από την πρώτη της Κομισιόν ε, όλη η περιοχή 6α ε, περιλαμβάνεται και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε και πρόσθετο αλίευμα, δηλαδή το 6α νότιο απόθεμα της Ρέγκας όμως ε, δεν ε, είναι ε, δυνατό να ρυθμίσουμε δύο αλιεύματα. Μας ενδιαφέρει εδώ με το σχέδιο να ρυθμίσουμε την περιοχή 6α βόρεια, 6 α North όμως, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι προθέση της Κομισιόν να προτείνει αύξηση στο πεδίο εφαρμογής ε, του ε, σχεδίου, αλλά να συνεχίσουμε τη διαχείριση του υφιστάμενου αποθέματος όπως και σήμερα. έτσι είναι τα πράγματα, δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξουμε τη διατύπωση, αλλά θα θέλει η Κομισιόν να μου αποσαφηνίσει και να μου βεβαιώσει ποια είναι η πρόθεσή της. Τώρα για το άρθρο 7. Αυτό το άρθρο έχει να κάνει με την αναθεώρηση των ποσοστών θρησιμότητας των ηχθείων και των ε, επιπέδων της βιομάζας. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν ήταν ε, πάρα πολύ αοριστή και δεν ανέφερε σε ποιες επιστημονικές αποδείξεις ε, βάσισαν τις τιμές. Εγώ θεώρησα τον απαραίτητο να βάλουμε διατύπωση ότι οι επιστημονικές συμβουλές θα πρέπει να έρχονται από το STECF και επίσης έχω βάλει και πλήρη διαβουλευσή με το Πελαγικό Περιφερειακό Γραμμοδοτικό Δημοτικό Συμβούλιο καθώς ε, το είχαμε στην αρχή στενή συνεργασία αυτού του Περιφερειακού Οικονομικού Συμβουλίου με το ISIS ε, πρέπει να τους συμπεριλάβουμε πλήρως και αυτούς τι μελλοντικέ διαβουλεύσεις και καθώς ε, είναι περιορισμένος ο χρόνος για την αναθεώρηση διατήρησα την πρόταση των κατεξουσιδότηση πράξεων διαδικασίες για να μην έχουμε καθυστερήσεις με την τακτική νομοθετική διαδικασία και στο άρθρο 8 τέλο σε συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν να προβεί σε streamlining της ε, αξιολόγησης ε, του σχεδίου και να έχουμε μία αξιολόγηση κάθε τέσσερα έτη και όχι ετησίως. Ε, έχω την εντύπωση ότι η το ετήσιο αίτημα για συμπαροχή συμβουλών ούτως ή άλλως δεν λαμβάνει χώρα και θεωρώ ότι η τετραετία, ακολουθώντας την τακτική νομική διαδικασία, είναι πιο κατάλληλη η Κομισιόν ε, θα πρέπει να ζητήσει ε, τη συμβουλή του Πελαγικού ΡΑΚ και του STCF, ε, όπως σας είπα, της, το και Νομίζω ότι έτσι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για τη διαδικασία. Ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Yes, uh, thank you. Ευχαριστώ να απαντήσω στις παρατηρήσεις του εισηγητού στο άρθρο 1. Πράγματι, θέλουμε να ρυθμίσουμε το ίδιο βιολογικό απόθεμο όπως τον παλιό κανονισμό. Καμία πρόθεση δεν υπάρχει να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, λοιπόν. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο? Όχι. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της μερσής διάταξης ελευτικέ δυνατότητε και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται συμφωνία ελευτική σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Μοζαμβίκη. Η κυρία Γκαρσία Γέρο έχει το λόγο για να μα παρουσιάσει το σχέδιο τη γνωμοδότηση που έχει αναλάβει. Παρακαλώ, κυρία Γκαρσία Γέρο. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Προσπαθούσα εδώ να τακτοποιήσω τα χαρτιά μου. Να σας πω ότι υπάρχει ένα λάθος στο κείμενο. Αντί για τη δεύτερη σελίδα, όπου γίνεται λόγος για 80.000 ε, τόνους, ε, γίνεται αναφορά σε 8.000. Είναι λάθος αυτό. και δυστυχώς έχει περισφρήσει στην ίδια την έκθεση. Όπως γνωρίζετε, το προηγούμενο πρωτόκολλο έληξε στις 31 ε, του 2011 και το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Κομισιόν για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις που κατόπιν ε, κάποιο χρονικό διαστήματος μας παρουσίασε τον Νοέμβριο πέρσι μας παρουσίασε μία έκθεση για να μπορέσουμε, σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες συναπόφασης που έχουμε, να θετήσουμε μία θέση θετική-αρνητική για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και το περιεχόμενό του. Μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση, γιατί η θέση ισχύ ήταν από την 1η Ιανουαρίου. Αλλά βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό δεν οφείλεται στις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ούτε είναι φταίξιμο της εισηγήτριας. Έτσι λοιπόν, ελαχθέντως αυτού, να πω τώρα κάτι σημαντικό. Οι πληροφορίες που θα έπρεπε να ε, συνοδεύουν ε, αυτή την έκθεση όπως ε, παραδείγματο χάρη, μελέτη περιβαλλοντικού δικτύπου και πιθανή περιβαλλοντική μελέτη. Δυστυχώς πριν να κάνω τη σύνταξη αυτής της έκθεσης δεν μπόρεσα να έχω στη διάθεσή μου αυτές τις πληροφορίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πληροφορίες που είναι στο δυνατόν πιο διαφανείς και να μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στο Κοινοβούλιο για να μπορείς κατόπιν να αρθρώσει μια πρόταση που θα πρέπει να είναι αντικειμενική και αληθής. Ε, γιατί διαφορετικά απλώς ε, λειτουργούμε με φορμαλιστικό τρόπο και δεν εκπροσωπούμε τους πολίτες. Τώρα, να αναφερθώ στο ίδιο το περιεχόμενο. Προτείνεται ένα νέο πρωτόκολλο που θα διαρκέσει τρία έτη από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Λοιπόν, κύριε Συνσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντισταθμίζεται στη συνέχεια μέσω αδειών που δίνονται ε, σε σκάφη που υλοποιούν την αλία. Στην Μοζαμβίκη έχουμε 980.000 ευρώ ετησίως, από τα οποία 530.000 ε, λεωμιλήτρια είναι αυτό που αφορούν την πρόσβαση των σκαφών ε, στην αλλιευτική ζώνη της Μοζαμβίκης και 400 70.000 έχουν να κάνουν με την υποστήριξη τομιακής πολιτικής για να βελτιωθεί ο τομέας της ελίας και η κατάσταση του πληθυσμού. Όπως σας είπα, έχουμε 8.000 ε, τόνους ε, ετησίω. Έχουμε μείωση σε σχέση με το προηγούμενο ε, πρωτόκολλο, 75 σκάφη συνολικά και έχουμε 43 αγριγροί και 32 παραγαδιάρικα επιφανείας. Κυρίες χώρες, ενδιαφέρονται είναι Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία. Οι νέε ε, τώρα ρήτρε που περιλαμβάνονται αφορούν κυρίω ε, την υποστήριξη του τομέα, ε, στην εργασία η Κομισιόν. Μάλλον η Επιτροπή Ανάπτυξης μας έστειλε μία σειρά συστάσεων και υποστηρίζει να εγκριθεί η έκθεση αυτή Απλώς ε, μας ε, επισημαίνουν ότι πρέπει ε, να φροντίσουμε να πληρούνται προποθέσει όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμός των δημοκρατικών ελευθεριών, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, να γίνονται σεβαστέ συστάσει του Διεθνούς Οργανισμού Εργασία. Όλε αυτέ τι συστάσει που, που πρέπει να συμπεριληφθούν ως νέε ρήτρε και θέλουμε ουσιαστικά να αποτελούν ε, μια ταυτότητα, ένα δελτίο ταυτότητας μέσω του οποίου τα δικά μας τα σκάφη και οι δικοί μας αλείς ε, ε, τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα προέλευσης και φυσικά θα ισχύουν και οι ίδιες συνθήκες ε, ε, και δεν μπορεί ποτέ ε, ο μισθός προηγούμενος χάρη του Νευτικού να είναι κατώτερος από ότι ο μισθός της χώρας της Ένωσης. Επίσης γίνεται λόγος σε αυτό το νέο πρωτόκολλο να πληρώνουν 20-25% περισσότερο οι εφοπλιστές και να φέρει την εγκαιότητα επιθεώρησης ελέγχου ε, και πρέπει με την Μοζαμβίκη να καθορίζουν σε ποια τοποθεσία θα γίνεται αυτή η επιθεώρηση. Και επίση ε, θεσπίζεται και ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίο για την καταγραφή όλων των δεδομένων που αφορούν τα ενέματα και ε, θα πρέπει να εγκριθεί από την 1η Ιουλίου και θα πρέπει να εμπλέκεται το Επιστημονικό Ινστιτούτο της Μοσαμβίκης. Εδώ γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης ε, και του ελέγχου των ελευτικών δραστηριοτήτων. Ε, από τη σκοπιά αυτή, όπως υπερασπίζουμε εδώ, θέλουμε μια βιώσιμη αλία και υπεύθυνη όχι μόνο στο ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκεί όπου ελεύουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλούμε για την εφορία όχι μόνο στη δική μας Ήπειρο, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Και έχουμε μία διπλή ευθύνη όταν εμείς πηγαίνουμε να λεύσουμε σε άλλες περιοχές. Γιατί θα πρέπει το όφελος ε, να δημιουργείται όχι μόνο και προς, ε, ναι, τον αφορά όχι μόνο τις χώρες και τα άτομα, αλλά θα πρέπει το όφελος ε, να είναι υπέρ και όλου του κλάδου. Έτσι λοιπόν, έχουμε και μία ρήτρα που λέει το εξής, στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι όροι, τότε μπορεί να υπάρξει ανάκληση, που μπορεί να είναι μερική, χρονική ή απόλυτη. Ανάκληση της άδειας. Και μιλώ για περιπτώσεις που δεν πληρούνται προϋποθέσεις, ε, είτε ε, στην περίπτωση που δεν έχουμε σεβασμό των ε, περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, είτε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε των δικαιωμάτων στον τομέα της εργασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας λέει ότι η ε, ε, διπλασιάζεται και η υποστήριξη στη Μοζαμβίκη με αυτή τη νέα συμφωνία και επίσης με θετικό τρόπο χαιρετίζεται σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση των δημοκρατικών αρχών των ανθρώπινων δικαιωμάτων να αναστέλλεται η άδεια, να ανακαλείται η άδεια. Και... Επίσης, ε, πρέπει να πούμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσοι αλλιεύουν στα της Μοζαμβίκης θα πρέπει να εφαρμόζουν όσο δυνατόν ε, μεγαλύτερη διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει γνώση των τεχνικών μέτρων που χρησιμοποιούνται για να υπάρχει καταπολέμηση της ε, παράνομης αλίας. Και επίσης ζητούμε να υπάρχουν αιτήσει εκθέσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας ε, και των πολιετών σχεδίων έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μία αξιολόγηση και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και μέτρα ανασύστασης του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορούν ε, να βελτιωθούν ε, να βελτιωθεί και οι συνθήκες αλίας αλλά και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της Μοζαμβίκης. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Ιέρο, η κυρία Λόφαν. Thank you very much, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρσία Χέρο Καραμπάλο. Είναι καλή η έκθεσή της. Συμφωνώ με την έμφαση που δίνεται στη διαφάνεια της προηγούμενης συμφωνίας. Η έκθεση αξιολόγηση πρέπει να διαβαστεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο εμπρόθεσμα κάθε φορά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρωτόκολλο με τη Μοζαμβίκη. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τις διαπραγματεύσεις αυτές τις πληροφορίες, γιατί αλλιώς ε, είναι αδύνατον. Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω, αλλά τι να κάνω. Ε, προετοίμαζα την συνεδρίαση και επειδή είμαι σκιώδης για τους πράσινους, για αυτή την έκθεση, ε, ήθελα να δω την έκθεση αξιολόγηση. Δεν πρόλαβα να πάω στη γραμματεία τη Αλία. Έπρεπε να υπογράψω, να πάω να δω την έκθεση. Δεν πρόλαβα, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι δημόσια αυτά τα έγγραφα ή τουλάχιστον να το λαμβάνουμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμείς ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, γιατί πώς να θέσω ευφύ αν δεν έχω ούτε καν τη σύνοψη της έκθεσης αξιολόγησης. Ευτυχώς η έκθεση της κυρίας Γκαρσία Γέρο Καραμπάλο είναι αρκετά πλήρης, όπως και η έκθεση Επιτροπής Ανάπτυξης. Αναφέρεται και ότι υπήρξε και έλλειψη διαφάνειας ως προς τις κοινέ συνεδριάσεις δύο επιτροπών. Πιστεύω ότι τα πρακτικά ε, θα πρέπει να είναι δημόσια όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το Κοινοβούλιο της Μοζαμβίκης. Ε, ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικρατεί διαφάνεια σε αυτές τις ε, αλληλευτικές συμφωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ένα-δύο πράγματα. Αναφερθήκατε στην αύξηση του, από το 20% στο 25% του τμήματος που πληρώνει ο πλειοκτήτης. Στη συνέχεια μιλάμε για 65 ευρώ τον τόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κανονική τιμή και γι' αυτό θέλω να ξέρω τελικά πόσα πληρώνει ο πλειοκτήτης ανατόνο βάσει της ε, νέας συμφωνίας. 300 ε, δολάρια το χρόνο αναφέρονται για το Ταμείο των ε, Εποπτών των Σκαφών. Μα είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσό. 300 ευρώ το ποσό είναι δυνατόν να ισχύει αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Πώς ε, χρηματοδοτείται η δράση των τοποτηρητών τώρα. Ε, τα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίου φυσικά είναι μια καλή ιδέα. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης με δορυφόρο VMS για τα... Υπάρχει πρόβλεψη να έχουν VMS ε, στο σκάφος τα... μιλώντας για τον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση πρέπει, όπως είπα, να διαβάζεται και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, αλλά και στο Κοινοβούλιο της Μοζαμβίκη. Η διαφάνεια θα πρέπει να επικρατήσει για όλους, όχι μόνο για μας. Ε, ε υποστηρίζω στην αρχή της αιρεσιμότητας. Αν υπάρξει παραβίαση, παραδείγματο χάρη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν δεν καταστήσει βιώσιμο τον κλάδο η Μοζαμβίκη, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αναστείλουμε την ε, ισχύ της ε, συμφωνίας να έχετε προβλέψει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε σχέση με αυτά που τονίζει η συγγήτρια της Επιτροπής Ανάπτυξης, ότι ανησυχεί για τη μη υποβολή των εκθέσεων αλλιευμάτων δυνάμει του πρωτοκόλου, όπως ε, αποκάλυψε η ex post αξιολόγηση που έγινε, Ωραία. Τι θα γίνει, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των πλειοκτήτων που δεν συμμορφώνονται. Ε, μόνο Ε, θα απειλούμε την Μοζαμβίκη με διακοπή της συμφωνίας αν δεν συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις. Εμείς αν δεν συμμορφωθούμε πώς θα ελέγξουμε τους πλειοκτήτες μας, πώς θα ελέγξουμε τη συμμόρφωση τους με τις διατάξεις της συμφωνίας. Ευχαριστούμε κύριο Στίβενσον τώρα. Ε, θα ήθελα... Να πω δύο λόγια κι εγώ για αυτά τα απόρριτα έγγραφα. Οι ευρωβουλευτές πρέπει να τα διαβάσουν αυτά, αλλά δεν μπορούν να, πάρουν, να κάνουν φωτοαντίγραφα, πρέπει να... Ούτε, πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να είναι παιδιά οι ευρωβουλευτές. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, σε ηλικία 10 ετών μπορεί να φέρνει λαθρέα ένας μεγαλύτερος το περιοδικό Playboy και έπρεπε να του δίνουμε, να τον ε, ε, χρηματοδοτούμε, να του δίνουμε ένα σελήνη για να μας αφήνει να δούμε τις φωτογραφίες. Ε, πώς είναι δυνατόν πάλι έτσι θα μας αντιμετωπίζουν εμάς τους ευρωβουλευτές. Είναι παράλογο πράγμα αυτό. Δεν είναι ότι περιμένει έξω από την πόρτα ο τύπος για να μας ε, πιέζει να δώσουμε αντίγραφο της συμφωνίας ε, σύμπραξης με τη Μοζαμβίκη. Δηλαδή είναι παράλογο το πώς χειρίζεται το θέμα η Κομισιόν. Η Κομισιόν και εγώ το ίδιο ήθελα να πω την ε, περασμένη εβδομάδα είχαμε λάβει και μια έκθεση από τη ΓΑΜΑ Εμπορίου. Ε, βέβαια υπήρχαν ε, κάποια έγγραφα που έπρεπε να παραχθούν και εκπονήθηκαν και υπήρχαν και κάποια αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν θέλω να παρακαλέσω την Κομισιόν, όπως λέει και ο κύριος Στίβενσον, να συνεχίσουμε να το διατηρούμε απόρριτο το θέμα αυτό του πλεμπόη, αλλά όχι τις εκθέσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν θα σχολιάσω το επεισόδιο περί Playboy, αλλά θα το διαβιβάσω στους ανωτέρους μου, ούτως ώστε να ε, αποδώσω πιστά τα όσα υπόθηκαν ε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ε, σχόλια εκτός μικροφώνου από την εισηγήτρια. Ε, θα ήθελα, συνεχίζει ο μιλητής, ε, να προσθέσω κάποια στοιχεία. Λοιπόν, για τις ε, αξιολογήσεις ανάμεσα πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Εντάξει, να επικρατήσει η διαφάνεια να είναι δημόσια τα έγγραφα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προφυλάξουμε κάποια απόρριτα στοιχεία για να μην γίνουμε όλοι ματάκιδες, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς πώς θα εφαρμόσουμε τη διαφάνεια για την έκθεση όταν ολοκληρώνεται υποβάλλεται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο οπότε κάνουμε ήδη μια προσπάθεια για να σας ενημερώνουμε καλύτερα ως προς την ε, ενδεχομένως ανεπαρκή χρηματοδότηση ε, σχετικά με τους, ε, το, εν πλώ. Ναι, όντω είναι χαμηλό το ποσό. Σας υπενθυμίζω βεβαίως ότι είναι το πρώτο πρωτόκολλο για τέτοιε συμφωνίε αλληλευτική ε, σύμπραξη. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, ένα σημείο εκκίνησης. Ε, το σημειώνουμε πάντω και όντω ίσω είναι υπερβολικά χαμηλό το ποσό. Τι γίνεται σε περίπτωση μη συμμόρφωση, υπάρχουν διάφορε διαδικασίε σε διάφορα επίπεδα. Πρώτον, ε, οι αρχέ ε, τη Μοζαμβίκη συζητούν το θέμα με στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής ή σε ε, ad hoc σύσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποτείνεται στο κράτος ε, σημαίας που, για το οποίο υπάρχουν υποψίες για την παραβίαση. Και το κράτος σημαίας, ως κράτος σημαίας αποφασίζει αν θα επιβάλλει ποινές στο σκάφος και θυμίζω ότι μπορούν και Καλά θα έκαναν ε, ε, οι αρχές της Μοζαμβίκης να μην ανανεώσουν απλώ την αλληλευτική δηλαδή άδεια ενό σκάβους που έχει κάνει μια παράβαση. Ε, ως ε, προς τα αιτήματα της Επιτροπής Ανάπτυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της σχετικές ρήτρε που υπάρχουν στη Συμφωνία, ε, φυσικά ε, θα το παρακολουθούμε και φυσικά η Μεκτή Επιτροπή θα κάνει απολογισμό σε συνεργασία με τις αρχές της Μοζαμβίκης ε, τακτικά σε σχέση με την υποστηρίξη της αεραστεχνικής αλίας, τις συλλογικές συμβάσεις και την ενίσχυση των μέσων ελέγχου. Με έχετε ήδη ακούσει για αυτό το θέμα και όπως είπε η συγγήτρια η τομεακή ε, στήριξη αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, ακριβώς μάλλον για να λειτουργήσει αισιότερα αυτός ο μηχανισμός. Τέλος, η εισηγήτρια τονίζει ότι χρειάζεται ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με τα άλλη επικαλυπτόμενα αποθέματα. Έχω και μια, ένα καλό νέο ε, να σας πω, δεν ξέρω αν είναι καλό το να, τέλος πάντων η Μοζαμβίκη ανήκει στο Συμβούλιο Τόνου του Ινδικού Ωκεανού πλέον. Ε, αυτό είναι ένα καλό νέο γιατί έτσι μπορούμε στην πράξη να εφαρμόσουμε ε, την ισότιμη μεταχείριση. Ευχαριστούμε κυρία Λεβίν. Μήπως θα μπορούσατε να δώσετε πληροφορίες κομισιών σχετικά με το ποσό που δίνουν οι πλειοκτήτες ανατόνων συγκεκριμένα. Και υπάρχει στη μοζανδική σύστημα VMS. Στο πλοία. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ από την Επιτροπή. Merci, Monsieur le Président. La réponse... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είναι ταχύ η απάντηση. 35 ευρώ τον τόνο. 35 ευρώ όπως και για τις υπόλοιπε εθιναλιευτικές συμφωνίες. Το VMS τώρα, το σύστημα παρακολουθήσης με δορυφόρο, από πέρσι είναι υποχρεωτικό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η συγκεντρία για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Προερχόμαστε από χώρες με διαφορετικές ε, διαδρομές. Έτσι λοιπόν δεν θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του κ. Στιβένσον ε, γιατί δεν αρμόζει. Και είμαι και γυναίκα, μην το ξεχνάτε. Εμείς ε, στην Ισπανία δεν μπορούσαμε να βρούμε τις πληροφορίες, δεν είχαμε πρόσβαση και δεν υπήρχε διαφάνεια, υπήρχε αδιαφάνεια, υπήρχε σιωπή και όλα αυτά μας έκανε να σκεφτούμε ότι ε, κάτι βρωμούσε. Ε, εγώ τώρα σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αναγνωρίσω ότι ε, κοιτάξτε, είπα θα είμαι και μόνο δύο μέρες μου έδωσαν ε, για να κάνω την παρουσίαση να τον κρίνουμε με επίγουσες διαδικασίε και να σταλεί και στη μετάφραση και σε όλους αυτούς και... μπορώ να σα πω ότι έλειπαν ορισμένα στοιχεία και ανέφερα και ορισμένου παράγοντε που έχει συμπεριλάβει η Κομισιόν που είναι πολύ σημαντική όμω. Ε, εγώ ε, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό είναι η, ε, περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου και κανείς δεν μου είπε πώς μπορούσε να έχω πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο και εγώ πήγα στην γραμματεία και δεν είναι η γραμματεία υπεύθυνη γιατί αυτό σε άλλο ε, πλαίσιο καθορίζεται. Και ήρθαμε στην Ισπανία, μα έλεγαν Να πηγαίνετε στο Υπουργείο να ψάξετε. Υπήρχαν τόνοι χαρτιά και δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πάρα πολύ εύκολο να ενημερωθεί κανεί για το πώ είχε η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για το θέμα που αφορά την διαφάνεια των πληροφοριών, λαμβάνοντα υπόψη και για το ότι ε, μας συστήνουν σε εμάς ε, ε τους ε, ε, βουλευτές ε, να ε, τα εξετάσουμε όλα αυτά και για, αυτό γιατί εκπροσωπούμε τους πολίτες και φυσικά εφόσον τέθηκε σε σκήση της Λαβώνας πρέπει να προσαρμοστούμε αλλά χρειαζόμαστε τώρα κάποια χρόνια για τη διαπραγμάτευση μια συμφωνία. δεν μπορούμε εμείς σε δύο μέρες ως κοινοβούλιο στη συνέχεια να δώσουμε μια θετική απόκριση για το θέμα αυτό. Τώρα εγώ εδώ κάνω αυτή την παρέμβαση γιατί με αποτέτουμε που να σας πω ε, δεν μου αρέσει ε, να βιάζομαι. Δεν ε, μου αρέσει να λειτουργώ γραφειοκρατικά. Δηλαδή, εμένα ε, με ενδιαφέρει όλα όσα λέμε εδώ να μην ε, μείνουν στη θεωρία και νομίζω ότι μεταξύ της ιδανοβλεψίας και της διαφάνειας υπάρχει μία ισορροπία, δηλαδή ότι πρέπει όσοι νόμιμα έχουν δικαίωμα να μάθουν τις πληροφορίες να τις μαθαίνουν και Τώρα, αν υπάρχουν κάποιε πληροφορίε που αφορούν ε, οικονομικέ ή κοινωνικέ πτυχέ, ε, δεν είναι πληροφορίε. Δεν είναι πληροφορίε αυτέ που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση του κράτου Μοζαμβίκη. Όμω, ε, από την πλευρά τη Κομισιόν, θεωρώ ότι υπήρχε καλή υποδοχή και νομίζω ότι το λάθο το έκανα εγώ, γιατί εγώ δεν γνώριζα ότι έπρεπε να κάνω το εξή και ζητώ συγγνώμη ότι έπρεπε να ε, ε, ζητήσω από την κυρία Λοβέ να κάνουμε μαζί ε, την έκθεση. Προσπάθησα να συμπεριλάβω ορισμένε πτυχές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πτυχές που αφορούν τους πόρους, για να πληρούνται. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που αυτά τα σκάφη λαμβάνουν κάποια ωφέλη, επειδή αλλιεύουν ορισμένα είδη με τα οποία έχω πρόβλημα βαθιά προβλήματα εκπεπιθήσεως. Ε, εγώ σας λέω ότι μπορούν να δοθούν περισσότεροι πόροι ακριβώς ε, έτσι ώστε να διευρυνθεί αυτός ε, ο φορέας της παρατήρησης. Εγώ νομίζω ότι για το μέλλον θα ήταν κατάλληλο να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, Εντάξει, ίσως ε, να δώσω έμφαση στο μέα κούλπα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, όμως ε, έμαθα τώρα και θα επιμείνω έτσι ώστε να φτάνουν σε εμά οι πληροφορίε γιατί ε, όταν διοριζόμαστε εισηγητέ, έχουμε δικαίωμα πρόσβαση στι πληροφορίε αυτέ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκαρσιαγέρο. Έχετε προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών μέχρι τις 2 ε, του μηνός το μεσημέρι. Τώρα, εδώ διακόπτουμε, θα συνεχίσουμε αύριο στις 3 το απόγευμα με την ε, συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και ε, να σας πω ότι δεν είναι σε αυτή την αίθουσα, είναι σε άλλη αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς στις 3. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο.